Um, so, um, let's, uh... Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίσουμε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Έχουμε ενημέρωση για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Άγκυρα, στην Τουρκία, 16 με 18 Μαρτίου που μας πέρασε. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Πρέντα να πάρει πρώτο το λόγο και μετά υπόλοιπη. Παρακαλώ κύριε Πρέντα πρέπει να συζητήσουμε τρία τέτοια θέματα. Δηλαδή σε λιγότερο από μία ώρα πρέπει να ενημερωθούμε για τρεις διαφορετικές ε, συνεδριάσεις, επισκέψεις που κάναμε ως Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα κάνω σύντομες παρατηρήσεις μετά από την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Άγκυρα. Πήγαμε υπό τον Έλμαρ Μπρόκ, τον πρόεδρό μας, δεν είναι εδώ σήμερα και γι' αυτό μου ζήτησε διακοπή από το ακροατήριο. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με την διερμηνία. Τώρα είναι εντάξει. Εντάξει. Κύριε Πρέντα, μπορείτε να συνεχίσετε. Έλεγα λοιπόν ότι στην αντιπροσωπεία μας ήταν μέλη από τις τέσσερις πιο μεγάλες πολιτικές ομάδες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι. Οχτώ ήταν τα μέλη της αντιπροσωπείας μας. Νετσμιάλη, εκ μέρους των Φιλελεύθερων, Αμιάτ Μπασίρ, εκ μέρους των Συντηρητικών, Κατυπήρη, εκ μέρους ε, των Φιλεύθερων που είναι συγητή του Κοινοβουλίου για την Τουρκία και άλλο ένας. Για το ΕΛΚ ο κύριο Μπροκ και εγώ ίδιο. Είχαμε και την κυρία Ζόμερ που είναι η εισηγήτρια και τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη ο οποίος είναι ο από κοινού πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μεικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Όσον αφορά τώρα τη συνάντηση αυτή καθεαυτή, έλαβε χώρα Τρίτη και Τετάρτη. Πολύ γεμάτες ήταν αυτές οι δύο μέρες με συναντήσεις αφενός με διάφορους υπουργούς, με Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό ή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων βέβαια, που είναι και αυτός που είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια μας είδε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Ερντογκάν και στη συνέχεια είχαμε και συναντήσεις με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων. Μας δόθηκε και η δυνατότητα υπό κατά κάποιο τρόπο. Υπό του βετριονά μας μπορέσαμε να συναντηθούμε και με δημοσιογράφους και με ακαδημαϊκούς κόσμο, δηλαδή από τους ακαδημαϊκούς και με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Οι συζητήσεις εκεί ήταν πολύ έντονες. Τώρα, τι θέματα είχαμε στην ημερήσια διάταξη. Θα τα αναφέρω, απλώς θα τα παριθμίσω. Δεν θα τα πω με τη σειρά. Με τι θέματα ασχοληθήκαμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, ασχοληθήκαμε με διάφορα κεφάλαια διαπραγματεύσεων. Εκφράσαμε την άποψή μας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και επίσης με τους Τούρκους συνομιλητές μας συζητήσαμε και για τη δυνατότητα ανοίγματο κι άλλων κεφαλαίων. Δόθηκαν διάφορα παραδείγματα τέτοιων κεφαλαίων. Αναφέρθηκαν τα 23 και 24, όπως επίσης και το 31, που έχει να κάνει με θέματα εξαταρκών υποθέσεων και ασφάλειας. Το 21 και το 24. Οι διαπραγματεύσεις TTIP επίσης μας απασχόλησαν. εκφράστηκε κάποια δυσαρέσκεια κατά κάποιο τρόπο από πλευρά των Τούρκων συνομιλητών μας που δεν είναι ενήμεροι για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Επ' αυτού εμείς συζητήσαμε επί μακρό και με προσώπους των Υπουργείων αλλά και κομμάτων το θέμα της ε, επαναδημιουργίας κατά κάποιο τρόπο της Θελωνιακής Ένωσης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί ω σύστημα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θίξαμε ήταν το θέμα της ενέργειας. Αναφερθήκαμε στον Ναμπούκο και εκεί είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από πλευράς της Τουρκίας που θέλουν συνεργασία και με εταίρους από την Ασία αλλά και Ευρωπαίους ακούσαμε την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί μας στον τομέα αυτών της ενέργειας. Ένα τέταρτο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν οι σχέσεις με την Αρμενία. Όπως γνωρίζετε το 2015 είναι ιδιαίτερη χρονιά όσον αφορά την μνήμη των ε, λαών του αρμενικού και του τουρκικού. Και κάποιος είπε, και το τονίζω αυτό, ότι πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο τουρκικών και αρμενικών ε, αρχών θα διευθετηθούν. Πιστεύω ότι τον Απρίλιο θα μας δοθεί ευκαιρία να συναντήσουμε μια αξιοπρεπή και σωστή αντιμετώπιση αυτού του τόσο ευαίσθητου θέματος. Πέμπτο θέμα, σχέσεις με τη Ρωσία. Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Διάφοροι Τούρκοι συνομιλητές μας γνωστοποίησαν ότι θα προτιμούσαν να είχαν ερωτηθεί πριν αποφασίσουμε για κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Κύπρος. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι καλώς συζητιέται τόσο πολύ στο Κοινοβουλίο, όμως δεν χρειάζεται εδώ να το τονίσω ιδιαίτερα και να σας εξηγήσω ποια είναι η θέση των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ποια είναι η θέση της Άγκαρας από αυτού, την ξέρετε, της από αυτού, τα ξέρετε. Άλλα θέματα τώρα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του καθεστώτος στην Τουρκία, το πολιτικό καθεστώς πρώτα απ' όλα. Συζητήθηκε η δυνατότητα αλλαγών μετά τις εκλογές δημοψήφισμα ή κοινοβουλευτική απόφαση. Όλα θα εξαρτηθούν από το συσχετισμό δυνάμεων που θα έχουμε μετά τις εκλογές. Ένα πάντως ιδιαίτερο σημείο ήταν οι εκλογές. Ήταν ακριβώς το ότι υπάρχει το 10% για είσοδο στο κοινοβούλιο και σε σχέση με αυτό υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που είναι η κατάσταση των Κούρδων και της εκπροσώπησής τους στη χώρα. Όπως γνωρίζετε, το Κουρδικό Κόμμα, το HSP, αποφάσισε να συμπεριληφθεί και αυτό στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο κόμμα και να μην ενσωματωθεί σε κάποιο άλλο κόμμα. Είχε 1,8% στις προεδρικές εκλογές, οπότε θέλουν να ξεπεράσουν αυτό και βέβαια υπάρχει πάντα κίνδυνος να μην ξεπεράσουν το όριο το οποίο προβλέπεται. Αυτό ήταν ένα θέμα λοιπόν που συζητήθηκε. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, συζητήσαμε και για την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία έκφρασης γενικότερα. Πολλές φορές αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι κλείσαν εκεί 600 σελίδες ε, στο, δια... στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η εκτίμηση τουλάχιστον των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τι οποίε μιλήσαμε. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα αυτό τη ελευθερία έκφραση και με του δημοσιογράφου και με άλλου. και είχαμε έντονε συζητήσει και όσον αφορά το καθεστώ των δημοσιογράφων στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε ε, για την έκθεση αντιπίδη που θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα στην Ολομέλεια. Οπότε θέλω να του δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, δηλαδή πρόεδρε, εφόσον συμφωνείτε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Η κυρία Πίδη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο. Δεν θα επαναλάβω τα όσα ήδη αναφέρθηκαν. Θα συμπληρώσω κάποια από αυτά. Για να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος, Κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι σχετίζεται με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε αυτό το κοινοβούλιο υιοθετήσαμε τον Ιανουάριο να ψηφίσουμε για την ελευθερία έκφραση μετά από τα όσα συνέβησαν το Δεκέμβριο και ακολούθησε η συζήτηση στην Τουρκία για το αντιφατικό ε, ε, σύνολο μέτρων για την ασφάλεια που ακόμα συζητείται στο Κοινοβούλιο. Τα μισά άρθρα έχουν ήδη υιοθετηθεί ενώ ενωμένοι η αντιπολίτευση και οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών θέτουν το ζήτημα ότι με αυτό το πακέτο για την ασφάλεια δίνεται υπερβολικά μεγάλη εξουσία στην αστυνομία παρακάμπτοντας το δικαστικό και φυσικά αυτό για μας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε σε όλες μας συζητήσεις με τους τόκους ομολόγους μας. Επίσης επαναλάβαμε αυτά που εδώ και μια πενταετία επαναλαμβάνει επικοδομητικά βέβαια το παρόν κοινοβούλιο και που θα συνεχίσει να λέει όσον αφορά εμένα ότι χρειαζόμαστε πιο εντατικό διάλογο επί αυτών των ζητημάτων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι ε, να κάνουμε έκκληση για να ανοίξει το κεφάλαιο 23 και 24. Και γενικότερα περισσότερο διαρθρωμένος διάλογος. Ε, σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτώντα τα όσα γίνονται νότια της Τουρκίας, στη Συρία και προς Ανατολάς, ε, χρειαζόμαστε έναν πιο διαρθρωμένο υψηλό επίπεδο διάλογο ε, για τις εξωτερικές υποθέσεις, το ίδιο και για την οικονομία. Ένα από τους συνομιλητές μας έδωσε το εξή παράδειγμα. Όταν εμεί ε, ρωτήσαμε τι διαρθρωμένο διάλογο υπάρχει τώρα για την οικονομία μα, είπε το εξή. Κάθε χρόνο μετά από τη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ, η Τουρκία όπω και άλλε υποψηφίε χώρε μπορεί να κάνει μια δεκαλύπτη παρουσίαση. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει όσον αφορά το διαρθρωμένο διάλογο. Ενώ γνωρίζουμε ότι ε, κάτι τέτοιο συμφέρει και εμά ε, με μεγάλο όγκο εμπορίου, το 70% των άμεσων επενδύσεων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε χρειάζεται περισσότερη δουλειά αυτό ο τομέα. Όπω ανέφερε και ο συνάδελφο, αναβάθμιση τη Ελληνική Ένωση, ε, εκφράστηκαν ανησυχίε από την Τουρκία ότι η τίτη μπορεί να έχει τρομακτικέ επιπτώσει όταν υπογραφεί η σύμβαση με τι ΗΠΑ ε, από την Ευρώπη μπορεί να έχει κάτι τέτοιο τεράστια επιπτώσει στην τουρκική οικονομία χωρί αυτή να έχουν ε, να πούν οποιαδήποτε άψη γι' αυτό. Για την ενέργεια και για την απελευθέρωση των θεωρήσεων επίσης. Τώρα όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, ε, αναγνωρίζουμε ότι παρότι ορισμένες φορές τα πράγματα δεν γίνονται όσο θα θέλαμε γρήγορα, πρέπει να δώσουμε επένους ε, στην τουρκική κυβέρνηση γιατί έχει δώσει φωνή μεγαλύτερη στους Κούρδους. Έχει βοηθήσει να προχωρήσει η διαδικασία κατά τη διαμονή μας όταν το HDP, το Κουρδικό Κόμμα, αποφάσισε να είναι υποψήφιο στις εκλογές της 7ης Ιουνίου, ακούστηκαν διάφορες, ε, διάφορα σενάρια για το κατά πόσο θα περάσει από αυτό το 10% αυτό το κατόφλιο και τι θα γίνει με την ενευτική διαδικασία ε, σε αμφότερες περιπτώσεις. Κατά τη διαμονή μας, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του HDP, του Κουρδικού Κόμματος, ο κ. Δεμεριτός, είπε σαφώς ότι δεν επιθυμεί να υποστηρίξει το AKP σε περίπτωση που δεν λάβει πλήρη, απόλυτη πλειοψηφία. Δεν θέλει να του υποστηρίξει για να δημιουργήσουν αυτή την υπερπροεδρία που θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα από κοινοβουλευτικό σύστημα σε προεδρικό σύστημα ώστε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό ζητήθηκε έντονα την περασμένη εβδομάδα εντό τη ίδια Τουρκία. Επίση αναφέρθηκαν και τα ζητήματα των προσφύγων και άλλο ένα ζήτημα το οποίο συχνά δεν τονίζουμε επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα αν δούμε την τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Τουρκία σε σχεδόν 2 εκατομμύρια Σύριους προσφύγους στην Τουρκία και πώς εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη και να συμβάλλουμε. Και κάτι τελευταίο, ένα από τα καλά αυτών των αντιπροσωπείων είναι όχι απλά ότι μπορούμε να εκφράσουμε, να διαβεβάσουμε τις ανησυχίες μας στους Τούρκους ομολόγους, αλλά και το αντίστροφο. Είμαι βέβαιη ότι θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε τις ανησυχίες των ομολόγων μας, όπως μας τις διαβίβασαν αυτοί. Κάτι που ακούμε κάθε χρόνο είναι ότι κατά την άποψή τους είναι άδικες οι διαδικασίες προσχώρησης. Θεωρούν ότι προσδιορίζονται περισσότερο πολιτικά παρά βάσει της αξίας τους. Τους ανησύχησε το ψήφισμα για το αρμενικό ζήτημα που θα ψηφίσουμε την 1η Ιουλίου και φυσικά το τελευταίο που είναι κάτι νέο είναι η Ισλαμοφοβία. Οι Τούρκοι ε, εξέφρασαν έντονες ανησυχίες. Μας είπαν δείτε τι γίνεται με τι ε, μουσουλμανικές κοινότητες ε, που ζουν στην Ευρώπη όσον αφορά θέματα, προβλήματα διακριτική μεταχείριση. Οπότε αυτά είναι ζητήματα που ακούσαμε εμεί από τους Τουρκου ομολόγου. Δεν σχετίζονται λοιπόν μόνο με τη διαδικασία ένταξης, αλλά γενικότερα με τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι Πολύ καλά. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ. Τάνοκ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κάποια θέματα θα ήθελα να αναφέρω και διαρωτώ με κάποιοι από τους συναδέλφους που πήγαν στην Άγκυρα αν μπορούν να απαντήσουν ή αν αναφέρθηκαν σε διμερείς επαφές. Ένα από τα ενηγματώδη θέματα διεθνώς είναι ποια είναι η συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και του Ισλαμικού κράτους Ιράκ και Συρίας και ποια προβλήματα τίθενται. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας πρόσφατα διέσωσαν στο Κομπανέ και κατάφεραν να διεισδύσουν σε ε, επικράτεια του οίκης... Διερωτώ με τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και τι τεκταίνεται. Διότι ε, αρνήθηκε με βάση το θέμα της εθνικής ασφάλειας να αποκαλύψει κάποια θέματα η Τουρκία για την Κύπρο, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την καταδίκη της θέσης της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά την δημοκρατία της Κύπρου και τα δικαιώματά της να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάνθρακες στα χωρικά ύδατα. Ε, δεν με εκκλείσει ότι σε σχέση ε, με την συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν βρίσκονται πολύ κοντά τώρα οι Τούρκοι με τους Ρώσους και σε σχέση και με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης εξάλλου. Αλλά εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι το γεγονός ότι η Τουρκία Τουρκία πάντα έλεγε ότι τα κλειστά σύνορα με την Αρμενία εξακολουθούν να υφίστανται λόγω του ε, αυτών που υφίστανται οι, Ισλαμισ... οι, οι μουσουλμάνοι αδερφοί στο Αζερμπαϊτζάν και σε σχέση με την χαζαρική ε, μειονότητα στην Κρυμαία που είναι, ε, βρισκόταν στην, ε, βρίσκεται στην ρωσική επικράτεια και έχουν εξοριστεί και μετά την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων όπου ε, μήμα ακριβώς ε, τη ε, της επαιτίου απότησης φόρου τιμής και μνήμης σε αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο και όπου συμμετείχαμε πρέπει να δούμε ακριβώς το τι γίνεται και τι γίνεται σχετικά με την Κρυμαία και το ΠΚΚ σε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση όπως είχε καταχωρηθεί και τις αλλαγές που έχουν ακολουθήσει σε σχέση με τις μάχες που δίνει το ΠΚΚ κατά του οίκης και εδώ σε σχέση και με τον Ατζαλάν διαρωτώ με, ανησυχούν οι Τούρκοι ότι ίσως σε σχέση με αυτήν την αλλαγή καθεστώτος υπάρχει κάποιο, κάποια νέα κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Εσείς παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν και εγώ, ήταν μια ερώτηση που και εγώ ήθελα να θέσω, λέει η κυρία Λούνατσεκ. Και τα άλλα δύο θέματα που θα ήθελα να ρωτήσω πιο εξειδικευμένα είναι, συναντήσατε και αν με συγχωρείτε αν μου διέφυγε, ζητώ συγγνώμη. Συναντηθήκατε με συλλόγους και ενώσεις δημοσιογράφων και γυναικών, διότι αυτά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά την Τουρκία σήμερα. Και το τι γίνεται με τον πρόεδρο Ερντογάν που έκανε λόγο για τον ρόλο των γυναικών και ότι θα πρέπει να περιορίζονται λέει οι γυναίκες ε, στο ρόλο τους στην οικογένεια και σε σχέση και με τις συλλήψεις δημοσιογράφων που βρίσκονται στις φυλακές. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ. Στεφαν Μπάλεν, Μπάλεν, παρακαλώ. Εξ ονόματος της Άντε, θα ήθελα να μας πείτε κάτι περισσότερο για το οι Τούρκοι που συναντήσατε, οι επίσημοι αξιωματούχοι, πώς βλέπουν τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι από εμά που συνάντησαν εκπροσώπους από την Τουρκία βλέπουν ότι υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον από τους Τούρκους για τις πραγματικές διαπραγματεύσεις και την εμβάθυνσή τους και λόγω των ε, προβλημάτων που υπάρχουν και σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης ίσως θα μπορούσατε να αναφέρετε τα σχετικά με το ενδιαφέρον των Τούρκων να γίνουν ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν αρκετές ερωτήσεις που έχουν σύλλεγει. Θα σας ζητούσα από τους δυο σας να απαντήσετε σύντομα σε αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Πρέντα θα ξεκινήσει και μετά θα συνεχίσετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με την ερώτηση της κυρίας Λούνατσεκ, ακριβώς γιατί η πολιτική της ομάδα δεν ήταν μαζί μας. Είμαι πεπισμένος ότι για τους φιλελεύθερους και τους συντηρητικούς έτσι καλλιώς θα πάρουν περισσότερες πληροφορίες από τα μέλη των ομάδων τους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή. Λοιπόν, όσον αφορά την, στις συναντήσεις που είχαμε με οργανώσεις για τις γυναίκες, δυστυχώς δεν είχαμε κάποια ειδική τέτοια συνάντηση. Χάσαμε μία συνάντηση με τον Chief Ombudsman για λόγους που έχουν να κάνουν καθαρά με τη διαχείριση του προγράμματός μας. Δεν ήταν θέμα πολιτικό. Όμως το θέμα των γυναικών τέθηκε σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τα πολιτικά κόμματα. Και στον έντονο αυτό διάλογο που είχαμε ανάμεσα στους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στις ίδιες συζητήσεις και δύο πλευρές. Οι δημοσιογράφοι να κατηγορούν για διάφορους περιορισμούς, για το πόσο έθραυστη είναι η κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και ακούσαμε και πολιτικούς, κυρίως από το ΑΚΑΠΕ, που επιχειρηματολογούσαν ότι αντίθετα το καθεστώς προσφέρει πλήρης ελευθερίες και ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης. Μας ανέφεραν διάφορα νούμερα μάλιστα. Ενώ τα άλλα πολιτικά κόμματα, όχι το ΑΚΠ δηλαδή, αλλά τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, θεωρούν ότι είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό. Για τον κύριο Φανμπάλεν τώρα, με δύο λόγια. Ίσως θα έπρεπε να το είχα πει νωρίτερα. Το κλίμα που επικρατούσε από πλευρά των συνομιλητών μας ήταν πολύ θετικό. Κάθε φορά αναφέρονταν σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν, και αυτό είναι μια έκπληξη, ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις διαπραγματεύσεις και όλο και μεγαλύτερη στήριξη μάλιστα για διάλογο όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά συζητήσαμε τα διάφορα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων και η γενική, το γενικό πνεύμα ήταν ότι πρέπει να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια για τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το ρώτησε ο κύριος Στάνοκ, όλα αυτά τα θέματα, ΠΚΚ κλπ, ISIS, αποκλειστική ζώνη Κύπρος, τέθηκαν και είμαι πεπισμένος ότι ο συνάδελφός σα, από την ομάδα σας δηλαδή που ήταν μαζί μας στην επίσκεψη αυτή, θα σας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Βεβαίως στηρίξαμε τις θέσεις που υποστηρίζει το κοινοβούλιο μας στα τρία ψηφίσματα που έχουμε εγκρίνει από την αρχή της θητείας μας μέχρι σήμερα. Από το 2009 μέχρι το 2014 εγκρίναμε δύο ψηφίσματα για την Τουρκία. Από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα, έχουμε γκρίνει τρία ψηφίσματα για την Τουρκία. Το περιεχόμενο των ψηφισμάτων αυτών υποστηρίξαμε. Αλλά είμαι πεπισμένο ότι και η κυρία Κατυπήρη από την πλευρά τη θα μπορέσει να συμπληρώσει τόσο σας είπα εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πύρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Κύπρο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη Πέραν από την ε, αντιπροσωπεία εξωτερικών υποθέσεων ε, μετά από δύο μέρες είχαμε μια συνάντηση του JPC οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν το βασικό θέμα που συζητήθηκε εκεί το θέσαμε και στην αντιπροσωπεία ΑΦΕΤ και φυσικά σε τελική ανάλυση όλοι θέλουμε να ξανακάτσουν στο διαπραγματευτικό τραπέζι και οι δύο πλευρές ε, της Κύπρου και ίσως να υπάρξει μια ευκαιρία τον Απρίλιο όπου τόσο η θα τελειώσει ε, η αποστολή της Τουρκίας τον Απριλίο και οι έρευνες επίσης θα ολοκληρωθούν τον Απριλίο από την εταιρεία που κάνει τις έρευνες νότια της Κύπρου. Οπότε ίσως να υπάρξει μια ευκαιρία μέσα στο επόμενο δίμηνο ή οι δύο διαπραγματευτικέ πλευρέ να ξανασυνεχίσουν να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση. Αυτό συζητήθηκε για τι κυρίω για τη Ρωσία. Φυσικά το συζητήσαμε. Είμαστε απόλυτα σαφεί σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο ότι είναι σημαντικό και οι υποψήφιες χώρες να είναι συμμαχοί μα σε τόσο, σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Να πω κάτι καλό που είδαμε από την τουρκική πλευρά, παρότι θα θέλαμε να είναι πιο δραστήρια, να μας υποστηρίζει πιο δραστήρια, την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος Ερντογάν ε, επισκεφθήκε την Ουκρανία, το είχε ανακοινώσει ήδη και σε εμά και έκανε μια πολύ σαφή δήλωση όσον αφορά τους Τατάρους της Κρυμαίας. Και υπήρξε κάποια δήλωση αλληλεγγύης για την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας. Ενώ ταυτόχρονα η Τουρκία ψήφισε στα Ηνωμένα Έθνη όταν έγινε ψηφοφορία για την καταδίκη της ε, παρανομής προσάρτησης της Κρυμαίας η Τουρκία ψήφισε όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. Για την Αρμενία φανταζόμαστε φυσικά ποιες είναι οι ανησυχίες ε, της τουρκικής πλευράς. Πρέπει όμως να πούμε ότι και το ζήτημα αυτό είναι τέτοιο που θα θέλαμε να γίνουν περισσότερα βήματα. Αλλά δεν μπορούμε να ε, μην παρατηρήσουμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Το να υπάρχει δηλαδή και η δυνατότητα να συζητηθεί το ζήτημα, να γίνονται διάφορα σεμινάρια σε πολλές πόλεις της Τουρκίας ε, όπου συμμετέχουν ε, ιστορικοί και ακαδημαϊκοί για να συζητήσουν το ζήτημα και επίσης έχουν γίνει και δηλώσεις. Πράγμα που δεν συνέβαινε τα περασμένα χρόνια. Ε, δηλώσεις και από τον Πρόεδρο και από τον Πρωθυπουργό. Μετά το ζήτημα για το ΠΚΚ και κατά πόσο έχει γίνει συζήτηση να βγουν από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν το θέσαμε ο ζήτημα, ούτε το έθιξε η τουρκική πλευρά γιατί συμφωνούμε όλοι ότι δεν αποτελεί θέμα της ε, ατζέντα που συζητάμε, είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Το PKK θα διοργανώσει μια συνάντηση τον Άνοιξη για να συζητήσει την πάυση των όπλων. Ξέρετε, αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά. Στην παρουσία στιγμή δεν ε, γίνεται ιδιαίτερα ενεργά δραστήρια μια τέτοια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Τουρκία. Κυρία Λούρατσεκ, ναι, φυσικά συναντηθήκαμε με δημοσιογράφους και είχαμε και μια διμερή συνάντηση με τον Ombudsman, με τον Διαμεσολαβητή, όπου συζητήσαμε τα ίδια θέματα. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος κατά τη συνάντηση JPC που έλαβε χώρα μέσα μετά τη συνάντηση με την ΑΦΕΤ, επίσης το συζήτησαν και συζήτησαν και με ενώσει των γυναικών και οι περιορισμοί στα μέσα μαζική ενημέρωση επίση αναφέρθηκαν πολλέ φορέ σε πολλέ συζητήσει και όπω είπα συναντηθήκαμε με τρεις δημοσιογράφους, έναν από την ομάδα Ζάμων, έναν από μια πιο κυβερνητική ομάδα, ο, ε, προκυβερνητικό όμιλο και έναν από την αγγλική έκδοση της Χωριέτα. Και όπως ξέρουμε όλοι εκπροσωπούν άλλη ομάδα αναγνωστών. Οπότε αυτό μας έδωσε μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία. Επίση πρέπει να πω φυσικά ότι και εμεί εκφράσαμε τι ανησυχίε μα. Κύριε Βαμπάλεν, πώ βλέπει η Τουρκία τη σχέση τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ίσω έκπληξη σε κάποιου από εμά εδώ. Αλλά ξέρετε, κοιτώντα τα προγράμματα υψηλού επίπεδου και ακούγοντα τι απόψει όχι μόνο των εκπροσώπων τη κυβέρνηση αλλά και όλων των κομμάτων τη αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα ουσιαστικά ότι για αυτού η διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πρώτη στι προτεραιότητέ του. Και επίση, ζητώντα και για άλλου ε, διαρθρωμένου διαλόγου υψηλού επίπεδου, κάθε φορά μα λένε ότι δεν πρόκειται να αποσύρουν και να σταματήσουν τι διαπραγματευτικέ ε, ομιλίε για την ένταξη. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε την πλειοψηφία του τουρκικού λαού, το 54% να είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μεταξύ των νέων ανθρώπων το ποσοστό αυτό είναι, ε, το, είναι τα δύο τρίτα. Τώρα το πότε η Τουρκία θα γίνει μέλος ε, και κατά πόσο θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολλοί κόσμοι έχει αμφιβολίες, γιατί όπως είδα αυτοί το βλέπουν ως μια διαδικασία η οποία είναι περισσότερο πολιτική παρά βασισμένη στην αξία τους. Έχουμε και άλλους δύο συναδέλφους που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Η κυρία Μαριαλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την ε, αντιπροσωπεία για το όσα έκανε εκεί και ακούγοντας τον κύριο Πρέντα και τους άλλους συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία, κατάλαβα ότι θέσατε τις ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση με το θέμα Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέσατε και ευαίσθητα ερωτήματα. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω εγώ, που ίσως να μην το κάνατε ακριβώς, ποιες ήταν οι αντιδράσεις των συνομιλητών σας στις ερωτήσεις σας. Δεν αμφιβάλλω ότι θέσατε τις σωστές ερωτήσεις όσον αφορά τη δικιά μας την ε, οπτική γωνία, αλλά θέλω να ξέρω ποια ήταν η αντίδραση των συνομιλητών σας, όπως το είπατε για τους δημοσιογράφους, οι άλλοι πώς αντέδρασαν. Θα ήταν πολύ σημαντικό για μας, ίσως όχι σήμερα γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά θα ήθελα να είχα ένα εγγραφό το οποίο να μου επιτρέπει να καταλάβω καλύτερα πώς βλέπουν τα πράγματα η υπεύθυνη από πλευρά Τουρκία. Αυτό θα μα βοηθούσε να καταλάβουμε ποια ακριβώ είναι η κατάσταση και τι δράσει θα έπρεπε να αναλάβουμε στο μέλλον στα πλαίσια των σχέσεών μα με την Τουρκία. Ευχαριστούμε, κύριο Μπασίρ. Πρόεδρο, και εγώ πήγα με την αντιπροσωπεία Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σε σχέση με το πώς είδα εγώ την, τις συναντήσεις αυτές. Παρά τις διάφορες παρεξηγήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες είχε σχέσεις με την Τουρκία. Σχέσεις από τις οποίες εποφελήθηκαν εκατομμύρια πολίτες εκατέρωθεν. Η Τουρκία σήμερα είναι ένας από τους δέκα πιο σημαντικούς εταίρους εξαγωγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια. Ανάπτυξη που δυστυχώς μόνο στον ύπνο τους θα μπορούσαν να, να δουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι προτιμούν επικεντρώνονται στα αρνητικά, ενώ εγώ πιστεύω ότι δεν επικεντρωνόμαστε αρκετά στα θετικά. Η Τουρκία ασφαλώς και πρέπει να φροντίσει να υπάρχει ένα καλό σύστημα δικαιοσύνης, ελευθερίας έκφρασης, κοινοβουλευτικού ελέγχου κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σημειώνουμε και που έχει επιτευχθεί πρόοδος. Έχουν γίνει πολλά βήματα για συμφιλίωση με τους Κούρδους. Η Τουρκία έχει κάπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία και ο νόμος, η νομοθεσία της για ε, τους ε, πρόσφυγες και το άσυλο είναι κάτι που τα ίδια τα Έθνη έχουν περιγράψει ως ε, πολύ θετικό που τηρεί τις αρχές κτλ. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το τελευταίο καιρό. Οικονομικά δε μιλώντας, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες στην ψηφιακή οικονομία της Τουρκίας. Η χώρα έχει 5 εκατομμύρια χρήστες ε, του διαδικτύου, πάρα πολλού στο facebook και είναι η 7 χώρα παγκοσμίως. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύει πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι υποδομές σίγουρα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να τις εκμεταλλευτούμε. Αν θέλουμε λοιπόν να βαθύνουμε στις στρατηγικές μας σχέσεις με την Τουρκία, ας προχωρήσουμε μαζί και σε επικεντρωθούμε στα θετικά. Η οικονομική ανάπτυξη και οι γερές διμερείς σχέσεις από το Δουβλίνο στην Άγκυρα θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και ευημερία για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Καστάλντο και μετά θα κλείσω τον ε, κατάλογο γιατί καταλαβαίνετε δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Όχι διμερός. Παρακαλώ κύριε Καστάλτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στους όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Θέλω να μου πείτε πιο συγκεκριμένα ε, περισσότερες προφορίες όσον αφορά το Turkish Stream, το γνωστό έργο που θα αντικαθιστούσε το South Stream συνδυάζοντας ε, στοιχεία ε, και του Ναμπούκο που ήταν ένα άλλο έργο το οποίο συζητήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου και ήθελα να μου πείτε κατά πόσο τέθηκε αυτό το θέμα στις διαπραγματεύσεις με τους ε, Τούρκους ομολόγους και τι θέση έχουν αυτοί όσον αφορά τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου έργου το οποίο αν δεν κάνω λάθος θα παίρναγε από την Ελλάδα, τη Φύρομ και τη Σερβία Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν ποιε ήταν οι δράσεις της Τουρκική πλευρά. Ευχαριστώ. Okay. <clears throat> So, I... Ωραία λοιπόν να σας ζητήσω να απαντήσετε στι ερωτήσεις είτε εσεί είτε κάτι γιατί πρέπει να συντομεύουμε. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Φυσικά με ευχαρίστηση διμερός μπορώ να συναντηθώ μαζί σας ε, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα σε σχέση με τους δημοσιογράφους ήταν μία από τις ερωτήσεις σας. Είναι η αυτολογοκρισία η οποία πολύ συχνά εφαρμόζεται από τους δημοσιογράφους τους ίδιους και προχωρούν και μέχρι του βαθμού της λογοκρισίας ε, στα κείμενά τους. Ένα από τα θέματα που θίξαμε είναι όταν υπάρχουν τέτοιες προσβολές ε, και ακούσαμε για περιπτώσεις στην Τουρκία όταν εκπρόσωποι της κυβέρνησης έχουν για παράδειγμα προσβληθεί από τα κοινωνικά μέσα και η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ως πολιτική αναφέρθηκε αν μας προσβάλλουν καθημερινά, αλλά αυτό ανήκει στη δουλειά μας ε, καθημερινά και αυτό ανήκει και στο πλαίσιο μιας ε, δημοκρατικής κοινωνίας, ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας, ότι μπορούν να εκφράζονται ελεύθεροι πολίτες εφόσον κάτι τέτοιο δεν ε, διώκεται και δεν μπορεί να τιμωρείται. Και για τα θέματα ασφάλειας και σε σχέση με την θέση της τουρκικής κυβέρνησης. Είδαμε το τι γίνεται και ποιες διατάξεις υπάρχουν και δεν υπάρχει ούτε μία διάταξη που να μην ε, υπάρχει σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας είπαν. Αλλά εμείς είπαμε ότι ιδιαίτερα με ένα τέτοιο μεγάλο, με τέτοια μεγάλη δέσμη για θέματα ασφάλειας οι Τούρκοι ίδια και με την προϊστορία, με την τρομοκρατία Γίνεται κατανοητό ότι είναι θέμα που ανησυχεί η ασφάλεια, αλλά ο σεβασμός των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπήρχαν διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την Επιτροπή Βενετίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε από τα δικά μας βιώματα και πείρα στην Ευρώπη να μπορούσαν να υποφεληθούν. Για τον κύριο Καστάλτο, για τα ενεργειακά θέματα και το τουρκικό, την τουρκική διαδρομή για το φυσικό αέριο ε, και τους ενεργειακούς πόρους. Συζητήσαμε σε σχέση με τους Τουρκούς ένα από τα πράγματα που ξέχασα να αναφέρουμε στην αρχή είναι ότι η επίσκεψή μας συνέπεσε με την ε, επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σεύκοβιτς που πήγε ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην Τουρκία ώστε να δοθεί το ανακτήριο λάκτισμα για τον ενεργειακό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για αυτά τα θέματα. Αυτά ήθελα να σας πω για, αυτό, αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Εσείς θέλατε να πείτε κάτι κύριε Πρέντα. Ε, Πολύ γρήγορα δύο σημεία. Οι διαφορετικές απόψεις ε, μεταξύ των Τούρκων είναι πολλές και διάφορες. Δεν υπάρχει ομοφωνία απόψεων και οι επικρίσεις αυτών προς εμάς είναι πολλές φορές ε, πιο λεπτές και πιο λεπτομερείς από τις δικές μας. Επίσης και τα δύο μέρη υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πολύ σημαντική συνεργασία τώρα με την Τουρκία δεδομένων των πολύ ευαίσθητων σχέσεων μας με τη Ρωσία και δεδομένων της κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κάποιος είπε μάλιστα σήμερα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο ενίσχυση των σχέσεων με την Τουρκία από ό,τι χρειαζόμασταν κατά τον ψυχρό πόλεμο. Αυτό χαρακτήρισε γενικώ τι τις ε, ανταλλαγέ απόψεων. Όπω και συναδελφό μου, φυσικά έχω να πω ότι είμαστε στη διάθεση των πολιτικών μας ομάδων για να δώσουμε περισσότερε προφορίες. Okay, thank you very... Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε αυτό το σημείο τώρα, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ. Και θα ήθελα να προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο, την ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη τη Αντιπροσωπεία Επιτροπή ΑΦΕΤ στο Ερμπίλ του Ιράκ και θα ζητήσω από τον κύριο Κάμ να μας κάνει μια παρουσίαση σε πέντε λεπτά, όχι περισσότερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από δύο συναδέλφους, εμένα και την ε, συναδέλφο Αγγιλάρα. Ο άλλος συναδέλφος ε, τα παράτησε δυστυχώς. Περάσαμε δύο μέρες στο Κουρδιστάν όπου συναντήσαμε σχεδόν όλους τους πολιτικούς ηγέτες πολλούς από τους μη κυβερνητικού οργανισμούς ε, και πολλές ομάδες που έχουν υποστεί επιπτώσεις από την κρίση και επίσης καταφέραμε να επισκεφθούμε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Θα είμαι σύντομο κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερις τομείς. Ο πρώτος αφορά τη μάχη κατά της ΕΝΤΑΣ, τη σχέση μεταξύ Ερμπίλ και της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης, την ανθρωπιστική κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος θέλω να αναφερθώ στο ευρύτερο πλαίσιο που κυριαρχεί στην περιφέρεια. Λοιπόν, το πρώτο, όσον αφορά τι μάχε, κατά σαφέ από την επίσκεψή μα ότι η παρέμβαση των διεθνών, της Διεθνής Συμμαχίας, της Διεθνούς Συμμαχίας έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα και ήτες στην ISIS. Αλλά πρέπει να πούμε ότι σε τελική ανάλυση απλά έχει περιοριστεί το ISIS, δεν έχει καταστραφεί λόγω τριών λόγων. Πρώτον, πολλοί μαχητές της ΔΑΣ είναι πρώην στρατηγοί υψηλά ιστάμενοι του ε, κόμματος Μπάθ ε, του Ιράκ που μετά τη διάλυση του δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά και έχασαν τις θέσεις τους ως ε, στρατιωτικοί. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εφάρμοσε διακριτική μεταχείριση κατά των Σουνιτών. Και ο τρίτος λόγος είναι το ISIS έχει, ε, παρότι έχει χάσει πολλά πυρομαχικά και όπλα, λαμβάνει όπλα από άλλους στρατούς που εγκατέλειψαν το πεδίο μάχης αφήνοντας τους τα όπλα τους και όπως και από τη Συρία επίσης ε, ε, λαμβάνει τα όπλα των, του στρατού του Ασάντ και ένας από τους συνομιλητές μας θεωρεί, μας είπε ότι εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 20.000 μαχητές. Ε, μας ζητήθηκε να παράσχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά γρήγορα στους Πέσμεργα ώστε να αναπτυχθούν ως δύναμη και το δεύτερο αίτημα ήταν να δούμε πώς θα γίνει η περιθάλψη των στρατιωτών στην Ευρώπη σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, έχει απαραίτητη τεχνολογία στο Ιρακικό Κουρδιστάν. Μετά τίθεται το ζήτημα της Μουσούλης και το ποιος θα πρέπει να ηγηθεί. Αλλά η δυσκολία είναι σαφώς ότι η Πεσμεργά δεν θέλουν να προβούν σε κάτι τέτοιο γιατί μπορεί να θεωρηθούν κατοχικές δυνάμεις ούτε οι επίσης. Ε. Οπότε όταν ε, τελικά θα αντιμετωπιστεί, θα επιληθεί το ζήτημα, το σημαντικό είναι να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Η πρώτη μας ε, σύσταση είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε να βρούμε μια συνολική λύση. Ε, έχουμε συζητήσει ήδη και με την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και πολλά ε, θέματα. Πρέπει να συζητήσουμε με τους ε, διάφορες ομάδες και η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τις δυνάμεις της ε, μπλοκάροντας ε, τη χρηματοδότηση προς το ISIS. Το δεύτερο θέμα είναι η σχέση μεταξύ Ερμπίλ και Βαγδάτης. Παρότι υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, παραμένουν δύο επίμαχα ζητήματα. Το πρώτο είναι η διένεξη για τα εδάφη και το δεύτερο ε, έχει να κάνει με το πετρελό και τα σχετικά έσοδα. Στα τέλη του έτους ε, παρουσιάστηκε λεπτομερώς αυτή η σχέση και το 17% ε, που χρησιμεύει για να τροφοδοτήσει την περιφερειακή κυβέρνηση που παρέχει πολλά δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση των Πεσμεργά. Παρά τη συμφωνία δεν έχουν διαβιβαστεί κονδύλια στους Πεσμεργά και αυτό έχει προκαλέσει σημαντικέ δυσκολίες στην κυβέρνηση εκεί, στην περιφερειακή κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ ε, ισχυρίζεται ότι έχει πρόβλημα ρευστότητας ε, και χρειάζεται το πετρέλαιο ε, περισσότερο από όσο τους διαβάζεται. Και οι Κούρδοι λένε ότι το 350 ήταν ο μέσος όρος και δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Ούτε οι δημόσιοι πάλι έχουν πληρωθεί, ούτε οι πεσμεργά έχουν πληρωθεί τα τελευταία χρόνια και Πέραν αυτών υπάρχει το όλο ζήτημα της κυβέρνησης της Βαγδάτης που δεν πληρώνει ουσιαστικά. Και υπάρχει και το πρόβλημα των προσφύγων. Να κλείσω με το προσφυγικό θέμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί πιέζει ο χρόνος. Ουσιαστικά υπάρχει τεράστια πίεση εκεί επισκεφθήκαμε τις περιοχές όπου υπάρχουν οι πρόσφυγες, συζητήσαμε με NGO επίσης. Κάπου όλοι λένε ότι υπάρχει ελευθερία κίνησης ε, και απασχόλησης αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη πίεση αυξήθηκε 28% ο πληθυσμό εντό εξαμήνου. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσει θα έχει αυτό σε οποιαδήποτε κοινωνία. Υπάρχει επίγουσα. Είναι αναγκαίο να βοηθήσουμε περισσότερο. Αφού τελειώσει και ο χειμώνα, αλλά ξέρετε, αυτό τελειώσει ο χειμώνα ε, οι θερμοκρασίε ανεβαίνουν στου 55 βαθμού, οπότε η κίνδυνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει εκεί μόλι φτάσει το καλοκαίρι. Οπότε χρειάζεται κάποιο επίγον σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση εκεί με κάποια χρηματοδότηση. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω με την τοπική εσύ και τι κυβερνήσει ώστε να αμβληθεί λίγο η πίεση εκεί. Θα σταματήσω εδώ και θα αναφερθώ στα υπόλοιπα ζητήματα όταν θα απαντώ σε ερωτήσει. Ε, ευχαριστώ κύριο Καστάλτο για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συναδέλφο κάνα για την πλήρη παρουσίαση του θέματος. έχω μια ερώτηση. Ωραία. Δεδομένου ότι είναι συμμερίζομαι και συμφωνώ μαζί του για να πολεμήσουμε την ΧΑΣ ε, αρκεί να βασιστούμε στη στρατιωτική επιλογή γιατί το να βοηθήσουμε πλήρως ε, υπάρχει και το πολιτισμικό, το οικονομικό πρόβλημα, το κοινωνικό το οποίο ε, είναι δύσκολο αυτό το θέμα της αρτολόγησης στη Δύση. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο συζητήσατε ε, τη σχέση μεταξύ ΔΑΕΣ και τα κράτη του Περσικού Κόλπου και την Τουρκία, ειδικότερα όσον αφορά όσον αφορά διάφορου ιδιώτε που χρηματοδοτούν το ISIS ε, μέσω διαφορών διάβλων και θέλω να πείτε αν μάθετε τίποτα όσον αφορά το παράνομο εμπόριο πετρελαίου δεδομένου ότι πριν από κάποιους μήνες ε, αναφέρθηκε ότι ίσω να εμπλέκονται και ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις και θέλω να μου πείτε κατά πόσο μάθετε τίποτα από του ε, ομολόγου μα στο Ερμπίλ. Επίση θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου όσον αφορά την αύξηση των χρηματοδοτήσεων για τους πρόσφυγες γιατί σίγουρα είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει από μόνο του το Ιρακινό Κουρδιστάν σε αυτή την ε, άνευ προηγουμένη αύξηση του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Καν. Λιγότερο από δύο λεπτά παρακαλώ. Συμφωνώ με αυτά που λένε οι συνάδελφοι στον Μπασίρ, αλλά για το δεύτερο, για το θέμα της Τουρκίας. Συζητήσαμε με διάφορους παράγοντες και όλοι έχουν την αίσθηση ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει περισσότερα. Και μερικοί μάλιστα λένε ότι η τουρκική κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο να βγάλει τον Ασάντα από την εξουσία παρά να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτος. για την ε, ιδιωτική χρηματοδότηση. Και εδώ θα έπρεπε να σταματήσουμε αυτή τη ροή. Πάντως δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να κάνει κάτι. Αυτά. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ τώρα. Δύο λεπτά. Σύντομα κι εγώ. Και μιλάω εδώ προσωπικά, όχι εκ μέρους της ομάδας μου. Ήμουνα και πρόεδρος της ομάδας φιλίας με το Κουρδιστάν που είναι διακομματική ομάδα. Κύριε Καν, δεν ξέρω αν το θέσατε ή αν συζητήθηκε τέλος πάντων το εξής. Το γεγονός ότι το KRG ήταν πρότυπο δημοκρατίας, σταθερότητας, μη θρησκευτικό, προστασία των μειονοτήτων, χριστιανών κλπ και άλλων, συζητήσατε καθόλου το σχέδιο δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση ή την ανεξαρτησία ως ανεξάρτητο κράτος. Ξέρετε από την ιστορία ότι οι Βρετανοί προσέφεραν ή αναγνώρισαν τέλο πάντων τη δυνατότητα δημιουργίας κουρδικού κράτους στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά έμεινε και σίγουρα είναι πολύ περίπλοκο το θέμα στα πλαίσια της κατάστασης που επικρατεί σήμερα και της ε, ομοσποδιακής δομής του Ιράκ. Πάντως, η ανακοίνωση του Προέδρου για δημοψήφισμα επ' αυτού είναι κάτι το οποίο συζητήσατε, καταλήξατε κάπου επ' αυτού. Ο κύριος Καν να απαντήσει. Ευχαριστώ και πάλι. Για το θέμα των μειονοτήτων. Το είπα και πριν. Πολλοί αναγνωρίζουν ότι είναι ανοιχτή η κυβέρνηση, ότι δέχεται διάφορα πράγματα. Είπαμε για ορισμένες περιπτώσεις η απάντηση είναι ότι πρόκειται μόνο για θέμα ελέγχου, τίποτα άλλο. Για τις μειονότητες συμφωνώ με αυτό που λέτε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στις σχέσεις με την κεντρική κυβέρνηση. Συμφωνώ. Για το δημοψήφισμα τώρα. Ναι, είχε σχεδιαστεί, αλλά εξαιτία Ισλαμικό κράτος η προτεραιότητά τους είναι να αντιμετωπίσουν αυτό το Ισλαμικό κράτος. αλλά βέβαια και τους ενδιαφέρει η ανεξαρτησία. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους πέρασαν πολλά δεινά. Τώρα το θέμα είναι να δούνε πώς θα λειτουργήσει κάποιο σύστημα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθούν με αυτό. πολλές από τις μειονοτικές κοινότητες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κεντρική κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα τα βρείτε και στην τελική μας έκθεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι ενημέρωση σχετικά με την τρίτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. 19 και 20 Μαρτίου. Ο κύριος Κούκαν, παρακαλώ, να μας ενημερώσει. Πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε προηγούμενα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμφωνία αυτή μεταξύ της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής που έγινε την προηγούμενη συνάντηση αυτή, την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή αν η δική μας αντιπροσωπεία ήταν η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία ΕΕ που επισκέφθη την Σερβία, 15 είμαστε εμείς και υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τους ε, βουλευτές μας για τις εξελίξεις της Σερβία. Στην αντιπροσωπεία μας υπήρχε και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού επίσης και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την μελέτη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης ε, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, Σερβία. Πήγαμε στο Νόβι Σαντ για να δούμε τη γέφυρα που κατασκευάζεται εκεί με αυτά τα κονδύλια. Το μεγαλύτερο αυτό σχέδιο, πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως προβλήματα που το συνοδεύουν. Η επίσκεψή μας στην περιοχή έδειξε και βοήθεια και απέδειξε στους ε, Σέρβους το ενδιαφέρον μας. Προτού ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε τη συνάντηση εργασίας με τους συναδέλφους από την Βουλή, την ε, Σκούπστινα, συναντήσαμε και τον κύριο Βούχσιτς και τον κύριο Σάσα Γιάνκοβιτς, ομπουτσμαν και τους εκπροσώπους επίσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτές οι συναντήσεις ήταν θα έλεγα συναντήσεις σε ένα πολύ ε, ειλικρινές και θετικό πλαίσιο. Και μέσα σε αυτές τις συναντήσεις, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, μπορέσαμε να εργαστούμε αποτελεσματικά. Υπήρχε μεγάλη βούληση να εκφραστεί η σοβαρή βούληση από πλευρά τη κυβέρνηση να προσεγγίσει η χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα. Αυτό προσπάθησαν να περάσουν ω μήνυμα και θα έλεγα και αρκετά πιστικά κιόλα τα κατάφεραν. Και σε σχέση και με τον Ombudsman, κάποιες ε, αναφορές είχαν ακουστεί ότι κάπως λέει υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με τη δράση του. Είδαμε ότι ο κύριος αυτός που είναι ο διαμεσολαβητής, ο Ombudsman, κάνει πολύ υπεύθυνα τη δουλειά του και αποτελεσματικά. Όσον αφορά το τώρα, μας είπαν ότι υπάρχει η πρόθεση να συνεχιστεί ο διάλογος ε, με τους εκπροσώπους του Κωσυφοπεδίου και ότι υπάρχει ανάγκη να επιληθεί το, το πρόβλημα του δικαστικού της δικαιοσύνης και το τι συμβαίνει με τους δήμους και κοινότητες εκεί. Η οικονομική μεταρρύθμιση που είχε προαναγγελθεί πέρσι τον Νοέμβριο έχει προχωρήσει πολύ καλά και έχει δώσει και καρπούς ε, για τους ε, κατοίκους και θα δούμε τι θα γίνει όταν θα εφαρμοστεί πλήρως η Σερβία διαδραματίζει ένα θετικό ρόλο στην περιφερειακή συνεργασία και για την σταθεροποίηση της περιοχής ε, διαδραματίζει θετικό ρόλο και μας διασφάλισαν ότι την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν και στο μέλλον. Όσο αφορά το κοσυφοπαίδιο θα έπρεπε να είχα προσθέσει ότι σήμερα υπάρχει μια δύο ημερών συνάντηση όσον αφορά την ε, ε, Πρίστινα, το κοσυφοπαίδιο σε σχέση με το βαλκανικό πλαίσιο. Έχει αποστείλει δύο εκπροσώπους η Σερβία και αυτό είναι μια ένδειξη ότι πιο ρεαλιστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα πλέον. Ενώ καμιά φορά λέγεται ότι ο διάλογος αυτός αυτό που κάνει είναι να πιέζει τη Σερβία, λέει, για να υπάρξουν οι παναχωρήσεις από τη Σερβία και ότι δεν είναι πραγματικός διάλογος. Βλέπουμε όμως ότι εδώ είναι δυνατόν ίσως να γίνει προσπάθεια να εξομαλυνθούν τα πράγματα και να υπάρξουν αποτελέσματα θετικά από αυτές τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Τώρα, η συνήθως, το συνήθως επώδυνο θέμα όσον αφορά την ε, υλοποίηση των κοινών συστάσεων ήταν αυτή τη φορά λίγο πιο δυνηρό και μας κάνει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσει να αναδιοργανωθεί το έργο αυτών των συνεδριάσεων στο πλαίσιο αυτό. Διότι υπάρχει πάντα πίεση χρόνου και αντί για συζήτηση ε, μιας ώρας ε, υπήρξε τριώρη συζήτηση, κόποση. Ένα άλλο πολύ προσωπικό θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η συζήτηση αυτή δείχνει ότι πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους, να συζητάμε μαζί τους πιο ανοιχτά, πιο ειλικρινά, σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε, ας το πω στην ίδια συχνότητα πολιτικού διαλόγου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ίδια αυτή, ας το πω έτσι, δυνατότητα συνεννόηση, στην ίδια συχνότητα. Υπάρχει υπερβολική ευαισθησία από πλευρά τους για κάποια θέματα και αντιδρούν υπερευαίσθητα και πρέπει να αποδείξουμε και να τους πείσουμε ότι είμαστε πραγματικοί φίλοι τους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε ειλικρινά. Θα έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια καλή επίσκεψη συνολικά αυτή και μάθαμε και κάτι καινούριο πώς να αντιμετωπίζουμε τους Σέρβους στο μέλλον. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Σερβία βρίσκεται στη σωστή πορεία, στη σωστή κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλά προβλήματα βέβαια που πρέπει να αντιμετωπίσουν αλλά και με πρόοδο που μπορεί να επιτελεστεί για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας της έκφρασης και θέματα που αφορούν την ίδια την κοινωνία. Όμως αν εφόσον προτίθεται να συνεχίσουν είμαστε εμείς ε, και εμείς διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε παρέχοντας υποστήριξη για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. No. Uh, Κύριο Κύριος όχι. Υπάρχει κάποιος άλλος. Κυρία Λούνατσεκ. Τον συνάδελφο Κούκαν που έκανε πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να υπάρξει και μια κοινή δήλωση στο τέλος τέλος. Θα ήθελα να προσθέσω δύο-τρία πράγματα για την αντιπροσωπή αυτή και για τη δική μου θέση. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κούκαν Πρέπει να έχουμε περισσότεροι, πιο ειλικρινείς ε, επαφές και διαλόγους μαζί τους. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, ένα θέμα. Οποιαδήποτε επίκριση ή κριτική ασκείται, οτιδήποτε αφορά κάποια, για παράδειγμα, δημόσια καταγγελία σε σχέση με τον Όμπουσμαν από κάποιους ε, ε πολιτικούς, ε, δεν ήταν δυνατό να δοθεί συνέχεια. Παρότι είχαμε κοινοβουλευτική συνάντηση δεν ήθελαν τα, οι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού να γίνουν τέτοιου είδους ε, δηλώσεις. Ε. Δεν, αυτό όμως είναι μέρος της ε, δημοκρατικής διαδικασίας και αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό και ενοχλητικό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα δημοκρατίας από πλευράς τους. Ένα πράγμα θα ήθελα επίσης να προσφέρω ότι και ακούσαμε από κάποιες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για παράδειγμα ότι μας είπαν ότι υπάρχει εντύπωση ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο, όχι από το Κοινοβούλιο, αλλά σε σχέση με το διάλογο για το Πέδιο, ότι αυτός λέει είναι ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμιά φορά θέματα για την ελευθερία των μέσων του τύπου και άλλα συναφή αμελούνται ή αγνοούν. Εμείς προσπαθήσαμε να τους πούμε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και τουλάχιστον αυτό το σημείωσα εγώ ως ε, μια παρατήρηση και για το θέμα του πώς οι σχέσεις διαμορφώνονται σε σχέση με τη Ρωσία σχετικά τουλάχιστον ο Πρωθυπουργό Βούτσιτς όταν μας υπενθύμησε ότι όταν επεσκέφθη ο Πούτιν τον Οκτώβριο νομίζω το Βελιγράδι ότι είπε δημόσια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προτεραιότητα για αυτούς αλλά και σε σχέση με την Σερβία κατά 95% εξαρτάται για τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων και καυσίμου, καυσίμων από τη Ρωσία η Σερβία. Και αυτό δεν είναι πολύ ισόρροπη η σχέση. Δηλαδή προτεραιότητα για την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τουλάχιστον όμως ε, για μας ε, δεν δίνεται η αναγκαία προτεραιότητα όπως θα το θέλαμε σε σχέση για τις σχέσεις με τη Ρωσία για παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει ο κύριος Πάσκου. Εντάξει. Ο κύριος Πιτουλά, λοιπόν, δύο λεπτά παρακαλώ. Και λιγότερο, πρόεδρε. Ένα λεπτό, λοιπόν, κύριε Πίκουλα. Για το Βελιγράδι θα ήθελα να προσθέσω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που είναι νομίζω σημαντικό αν θέλουμε να σταθμίσουμε και αξιολογήσουμε σωστά τι, συνέβη στο, τι έχει συμβεί στο Βελιγράδι. Είναι η μη ε, υπαρκτή συνεισφορά από πλευράς της σερβικής αντιπολίτευσης και κατά τη διάρκεια της συνάντησης ή της ε, ε, ίδιας της διεξαγωγής στο Κοινοβούλιο και την προσπάθεια να υπάρξει αναζήτηση κοινών συστάσεων τίποτα δεν ακούστηκε από πλευράς της αντιπολίτευσης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή της σημερινής πολιτικής κατάστασης και ζωής ε, στην ε, Σερβία. Και σε σχέση με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ που θίξαμε το θέμα μαζί τους κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το μεσημερινό γεύμα μας είπαν ότι αυτό δεν είναι καθόλου ε, θετικό και είναι μια νοσηρή κατάσταση και ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία και δραστηριοποίηση από πλευρά τη αντιπολίτευση. Θέλω να εκφράσω λοιπόν τη θλίψη μου, την απογοήτευσή μου για το ότι σε σχέση με τους, την πλειοψηφία των συναδέφων από τη σερβική πλευρά αρνήθηκαν έστω και μία ε, επίκριση ή κριτική όταν ε, στόχευε στην αναφορά κάποιων προβλημάτων όσον αφορά για παράδειγμα τα μέσα ενημέρωσης, ε, τα κοινωνικά μέσα, τον ρόλο του Ombudsman και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Φυσικά στη συζήτηση για την συνεισφορά των Σέρβων στην περιφερική συνεργασία. Εντάξει, αυτό συζητήθηκε, αλλά δεν επαρκεί νομίζω, διότι η περιφερική συνεργασία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας είναι κοινό στόχος και θα θέλαμε να δούμε να είναι πιο ανοιχτή σε σχέση με τέτοια θέματα και παρεμβάσεις οι Σέρβοι ομόλογοι μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ ο κύριος Πλένκοβιτς παρακαλώ. Ζήτησε να του επιτραπεί να κάνει μια σύντομη παρουσίαση σε σχέση με την συνάντηση της Ολομέλειας σε σχέση με την Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα. Ζητώ λοιπόν να μας ενημερώσει σχετικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αναφέροντας λέει ο κ. Πλέγκοβιτς ε, το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τις δραστηριότητες στο επίπεδο εξωτερικών σχέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι οι 25 ευρωβουλευτές συμμετείχαν στη Euronest σε σχέση και με το Γερεβάνο που ήταν μια, ένα πολυσχηδές εγχείρημα. Υιοθετήθηκαν δύο ψηφίσματα όσον αφορά την ε, δράση της Ρωσίας ε, στην Ουκρανία και την προσπάθεια να υπάρξει επίλυση του προβλήματος, την ε, γενοκτονία των Αρμενίων, ένα πολιτικού χαρακτήρα και ένα ενεργειακού πολιτικού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό το τελικό μήνυμα της Euronest κοινοβουλευτικά θα συμφωνηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι θα δοθεί ένα σαφές μήνυμα για τα όσα τεκταίνονται και βρίσκονται υπό εξέλιξη. Ο κύριος Σαρκασιάν, Αρμένο, πρόεδρος της Αρμενίας, δεν ήρθε ο εκπρόσωπος των Αζέρων στη, στο Γερεβάν. Υπήρξαν άτυπες συναντήσεις ε, με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της Μπελαρούς και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σημαντικό ότι υπήρξε και η συμμετοχή του Επιτρόπου Χάν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλη παρατήρησή μου, αν συμφωνείτε κύριε Πάσκο να αναφερθώ σε δύο παράλληλες ε, ε, ε, δράσεις. Η κυρία Φωτίγα για παράδειγμα και για την Επιτροπή Προϋπολογισμών που συναντήθηκε στο Κίεβο με την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας και δείχθηκε, καταδείχθηκε η συνεκτικότητα της κοινοβουλευτικής προσπάθειας με την παρουσία και της, ε, τη συμμετοχή των ε, υψηλών αξιωματούχων. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία Μίνσκ για την ειρήνευση και πώς ε, αντιμετωπίζεται το θέμα της αποκέντρωσης των περιφερειών αυτών υπό τον όρο να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες τίμιες εκλογές καθώς επίσης και τη νέα ημερήσια διάταξη που έχει υιοθετηθεί την προηγούμενη Δευτέρα από πλευράς του Συμβουλίου για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Και αρκετοί πολιτικοί από πλευράς της ε, Ουκρανίας συμμετείχαν και το θέμα των προσφύγων και η επίσκεψη στο Μαϊντάν. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί λοιπόν αυτός ο διάλογος. Από τους συναδέλφους μας, ε, με τη Βερχόβνα Ράντα, την Άνω Βουλή δηλαδή, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτές τις επαφές, ε, να συνεχιστεί η προσπάθεια σε σχέση με την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στην έκθεση για την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Μετά θα ψηφίσουμε. Δεν θα σας διαβάσω τα πάντα σε σχέση με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, αλλά θα ζητήσω από τον εισηγητή μας, τον κύριο Καμπριέλιους Λαντσμπέργης, σε πέντε λεπτά να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα. Και μετά δύο λεπτά θα έχουν το χρόνο οι ευρωβουλευτές να σχολιάσουν, να ρωτήσουν κλπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε έχω την αίσθηση ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις που εξετάζει αυτή την εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου το ενδιαφέροντος που έδειξαν οι συνάδελφοι όταν άρχισα να συντάσω την έκθεσή μου αυτή. Και όσο φτάνουμε πιο κοντά στην ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα τον Ιούνιο στην Ολομέλεια, τότε θα δούμε το ενδιαφέρον να αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Ας αρχίσω λιγάκι από τη διαδικασία που ακολούθησα. Λοιπόν, εδώ και πέντε μήνες περίπου δουλεύω πάνω στην έκθεση αυτή. Έχω συναντηθεί με όλους τους σκιώδεις συζητητές των πολιτικών ομάδων με τους οποίους είχαμε πολύ καρποφόρες συζητήσεις. Ανταλλάξαμε απόψεις για τη μορφή πρώτα απ' όλα που πρέπει να πάρει η έκθεσή μας. Συναντήθηκα και με εκπροσώπους από διάφορα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί πρέπει να πω ότι διαφέρουν μεταξύ τους κατά πολύ. Όταν βγεις από το γραφείο σου και πας στις διάφορες διευθύνσεις, θα διαπιστώσεις ότι έχουν διαφορετικές απόψεις για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία η αντιπροσωπεία μου έπρεπε να πάει στη Ρωσία, να βρεθεί όχι μόνο με τους αξιωματούχους στη Ρωσία, αλλά να συναντηθεί και με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά πρόκυψε θέμα με τις θεωρήσεις και δεν μπορέσαμε τελικά να ακούσουμε τις απόψεις όλων αυτών. Όμως, μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω με τον κύριο Πουσκόφ όταν αυτός ήρθε στο Στρασβούργο και του παρουσίασα την άποψή μου και να τι μου είπε. Δυστυχώς, τίποτα καινούριο δεν υπόθηκε, πέρα από αυτά που ακούμε συνήθως από τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. Βέβαια, κάποιες αποχρώσεις θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει για την ανάμειξη της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν το θέμα ετίθετο ξανά και ξανά. Τώρα θα περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων με τους κοιόδης εισηγητέ και όποιον άλλον ευρωβουλευτή ενδιαφέρεται για να ετοιμάσουμε τις τροπολογίες. Για να επανέλθω πάντως στο κείμενο. Όταν ε, άρχισα με την έκθεση αυτή, μου είπαν ότι κάτι που θα έπρεπε να αποφύγω στην έκθεση είναι να ακολουθήσω τον τίτλο. Και υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να το κάνω. Τώρα όμως, πέντε μήνες αργότερα, ε, είναι δύσκολο. Και δεν φταίω εγώ. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαίνει ότι όλοι είμαστε θύματα των τίτλων, των μέσων ενημέρωσης, όχι του τίτλου των ε, νέων που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης. Άμα βλέπουμε ότι αποσύρονται τα τάγκς, ότι δεν σκοτώνεται ο κόσμος κτλ, επικριτικά σχολιάζουμε θέλουμε να προχωρήσουμε για να συνεχίσουμε μετά όπως πριν. Αν όμως δούμε ότι γίνονται βομβαρδισμοί, ο κόσμος πεθαίνει, τότε ζητάμε ένα πιο σκληρό κείμενο και θέλουμε πιο αποφασικά μέτρα να ληφθούν σε βάρος της Ρωσίας. Επιδεζόμαστε δηλαδή από τους τίτλους των εφημερίδων. Και είναι αδύνατο να ακολουθήσουμε μία στρατηγική για πέντε χρόνια, ούτε καν για ένα χρόνο εφόσον δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση. Αν ξέρουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, ναι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας αναφέρω κάποια θέματα που θέλω να περιλάβω στην έκθεσή μου, πέρα από τους τίτλους των εφημερίδων. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια μοναδική ευκαιρία τώρα να αντικατοπτρίσει στην έκθεση αυτή την κατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία. Το 2012 ήταν πιο δύσκολο, το 2008 ακόμα πιο δύσκολο με την Γεωργία, για παράδειγμα την επίθεση στη Γεωργία. Τώρα όμως έχουμε όλοι τη δυνατότητα να πούμε ότι έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Είναι κάποιες κόκκινες γραμμές που έχει περάσει η Ρωσία και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν μπορούμε πια να πούμε ότι θα συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το άλλο είναι ότι πρέπει να αναφέρουμε πως είναι στο, στα χέρια της Ρωσίας να κάνει κάτι για να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη μας. Υπάρχει το Μίσκ 1, υπάρχει το Μίσκ 2, αλλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι μόνο οι συμφωνίες του Μίνσκ 2 που πρέπει να τηρηθούν. Είναι το θέμα της Κρυμαίας, είναι το θέμα της ενέργειας. Πριν την κρίση στην Ουκρανία υπήρχαν εμπορικοί πόλεμοι, και πολλά πράγματα τα οποία έπληταν και ε, ουσιαστικά έπληταν την εμπιστοσύνη που είχαμε στη Ρωσία. Τι βγαίνει τώρα από αυτή την κρίση. Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να βγει από αυτή την κατάσταση περισσότερο ισχυρή και περισσότερο ενωμένη. Και φαίνεται αυτό. Κάθε φορά που ψηφίζουμε στην Ολομέλεια έχουμε 500 περίπου βουλευτές που ψηφίζουν υπέρ των ψηφισμάτων για την Ουκρανία και στην τελευταία ολομέλεια. Είμαστε ενωμένοι. Και το 2008 ή και πριν από δύο χρόνια ακόμα θα ήταν πιο δύσκολο να περάσουν με τέτοια πλειοψηφία αυτά τα ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να δείξει ότι είναι πιο ανθεκτική και το τονίζω αυτό. Και θέλω να παραμείνει ο όρος αυτός resilient στην έκθεσή μου. Απέναντι στην προπαγάνδα, απέναντι στους εμπορικούς πολέμους, το πόλεμο για την ενέργεια κτλ. Τι μπορούμε να αντισταθούμε καλύτερα. Κάτι ακόμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανοιχτή. Θα παραμείνει ανοιχτή στο διάλογο, ανοιχτή στη διπλωματία, εάν η Ρωσία μάθει το μαθημά της αν καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη μας απέναντί της. Θα παραμείνουμε ανοιχτοί στους ανθρώπους, στον κόσμο, σε φοιτητέ που θα έρχονται στην Ευρώπη. Θα παραμείνουμε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή κοινότητα. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που βοηθήσατε να ετοιμάσω το σχέδιο έκθεσης που έχετε μπροστά σας. Να ξέρετε ότι θα παραμείνω σε επαφή μαζί σας και όσο προχωράει ο χρόνος και πλησιάζουμε στην ψηφοφορία, να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουν ζητήσει το λόγο διάφοροι συνάδελφοι και σκιώδεις που βρίσκονται εδώ παρόντες. Συνεπώς, δύο λεπτό καθένας το πολύ, παρακαλώ. Αλλιώς, μετέχουμε και μια κοινή συνεδρίαση με τους συναδέρφους από την Επιτροπή Πολιτισμών, οπότε μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Πρέντα πρώτα, για δύο λεπτά παρακαλώ κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συναδελφό, τον συναδελφό Λαντσπέργης. Η έκθεση του είναι εξαιρετική όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας το κείμενο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι υπογραμμίζει πολύ καλά την εξέλιξη των σχέσεων μας ε, με τη Ρωσία. Και δείχνει ποιες ήταν ε, κατά καιρός οι θέσεις της Ένωσης ε, και ποια είναι η σημερινή θέση. Το γεγονό ότι πλέον η Ρωσία δεν είναι στρατηγικός εταίρος της Ένωσης, ούτε πρόκειται να υπάρξει εάν δεν σεβαστεί τις διεθνείς συμβάσεις και τα σύνορα των ε, γειτόνων μας. Όπως έχει υποθεί επανελειμμένος, είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τη Ρωσία, αλλά σε καμία περίπτωση υπό τις τωρινές συνθήκες. Για να συνεργαστούμε, η Ρωσία έχει να κάνει πολύ δρόμο για το σεβασμό της παγκοσμίας τάξης, ε, της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των γειτόνων της. Ταυτόχρονα πιστεύω πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις θέσεις ε, που έχουμε υιοθετήσει ήδη. Χαιρετίζω έτσι την αποφάση του Συμβουλίου το, στο τέλος περασμένης εβδομάδας να συνδέσει τις ε, κυρώσεις ε, με τις ε, ε υπόλοιπες συμφωνίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα διότι καθημερινά βλέπουμε ότι οι συμφωνίες ε, που υπάρχουν ε, δεν ε, γίνονται σεβαστές από τη Ρωσία. Και όλοι έχουμε συμμετεί στην εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κρυμαία. Σε μερικές μέρες θα κλείσει ένα έτος από την προσάρτηση της Κρυμαίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρος. Η κυρία Γιακονσάρη, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω φινλανδικά λοιπόν. Και εγώ θα ήθελα τον Γκαμπριέλης Λαντσμπέργης να τον συγχαρώ για αυτή την έκθεση σε σχέση με τις, ε, όσο αφορά τις σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας. Έχει μια λογική δομή η έκθεση. Όμως το όραμα, η προοπτική είναι αυτό που χρειάζεται και να δούμε και την φιλοσοφία. Το ότι όλα δηλαδή τώρα εξαρτώνται λέει από τη Ρωσία. Αυτό δεν το βρίσκω κάτι το χαρακτηριστικό για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να υπάρχουν σειράξεις. Ούτε θέλουμε να ταπεινώσουμε φυσικά ή να ευτελίσουμε τη Ρωσία. Είναι σαφές βέβαια ότι υπάρχει προϋπόθεση εδώ ότι θα επιληθεί η κρίση στην Ουκρανία για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Και η εξομάλυνση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη συμφωνία του μη του Μίνσκ, της Λευκορωσίας. Θέλουμε λοιπόν με επικριτικό πνεύμα να αντιμετωπιστεί το θέμα της Ρωσίας. Έχουμε πολλές εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και έχουμε και πολλά ψηφίσματα που εγκρίναμε που αφορούν τη Ρωσία. Η Ρωσία η ίδια παρέβει, παραβίασε το διεθνές δίκαιο και εμείς αντιδράσαμε, υποχρεωθήκαμε να αντιδράσουμε. Η ενότητα και η ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική υπόθεση έναντι της Ρωσίας εκφράζουμε αυτή την επίκριση, την κριτική στάση που εκφράζουμε. Όσον αφορά όμως θέσεις ακραίες ε, ε, κάποιων ε, που θεωρούν ότι σε σχέση με την ενότητα η οποία θρηματίζεται λέει ή διαβρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υιοθετήσουμε ακραίες επικρίσεις ή να επαναλάβουμε τέτοιου είδους ακραίες θέσεις. Η συνεργασία θα πρέπει να ε, αποτελέσει θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα μην έχουμε αυταπάτες όσον αφορά τη Ρωσία αναφέρθηκε ότι εδώ δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε όπως και παλαιότερα λες και τίποτα δεν συνέβη business as usual δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο αλλά σε σχέση με την έκθεση όπου κάποιες φωνές ακούγονται δηλαδή εγώ βλέπω ότι λείπει η παγκόσμια προοπτική τα ε, θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου για παράδειγμα μέσα σε αυτή την προοπτική και το θέμα των λεσβίων και ομοφιλοφίλων που διώκονται και είναι αντικείμενο ε, διώξεων καθώς επίσης και να δούμε τις ε, εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν χωρίς να έχουμε αυτά πάτες για τη Ρωσία. Λυπούμε που είναι περιορισμένος ο χρόνος να παρέμβω, πολλά θα ήθελα να πω. Φωτίγα, δύο λεπτά παρακαλώ. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η κοινή προσπάθεια και συντονισμένη προσπάθεια και χάρη στο έργο του κυρίου Λαντσμπέργης, χάρη σε όλη αυτή την προσπάθεια μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Αυτή η έκθεση έχει κέρια σημασία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ όμως από την άλλη πλευρά παρόλα αυτά, παρόλη τη βούληση αυτό το έγγραφο να έχει οικουμενικότητα ή οικουμενικό χαρακτήρα αν θέλετε πρέπει να υπάρξει αναφορά και να τοποθετηθούμε σε πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται στην καθημερινή τους ε, ε, έκφραση σε σχέση με τη Ρωσία. Θα ήθελα περισσότερα τέτοια γεγονότα να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν ή να σταματήσουν την ε, Ρωσική Ομοσπονδία στην πορεία που ακολουθεί. Σε σχέση δηλαδή με την λογική που διέπει την Ρωσική Ομοσπονδία. Ο κύριος Μπορίς Νεμτσόφ δολοφονήθηκε. Και αυτό γιατί. Επειδή συμμετείχε ακριβώς σε σχέση με το έργο συνεργασίας που είχε αναπτύξει με τη διεθνή κοινότητα. Ήταν υπέρ των κυρώσεων που θα έπρεπε να επιβληθούν σε κάποιους εκπροσώπους της Ρωσίας και αυτή ήταν η αντίδραση τελικά σε σχέση με την ε, προσάρτηση από την Ρωσία της ε, ε, Κρυμαίας και ρόλος ήταν να ενταχθούν περισσότερα ονόματα υψηλών αξιωματούχων στο μαυροπίνακα, στην λίστα δηλαδή των Αμερικανών που ε, θα συμπεριλάμβανε αυτά τα άτομα. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν πρέπει να αναλυθούν και να, αναλυθούν και να ληφθούν υπόψη ως γεγονότα και σε αυτή την έκθεση. Τέτοιου είδου στοιχεία δηλαδή. Η Ουκρανοί εταίροι μας από την άλλη πλευρά προσπαθούν και εκείνοι να είναι πολιτικά ορθοί εντό εισαγωγικών. Υιοθετούν και διέπονται από την ίδια λογική όπως και εμείς θέλουν να ε, κατευθύνονται και να προσανατολίζονται με τους όρους της συμφωνίας ε, του Μίνσκ και θα ήθελαν οι κυρώσεις να είναι πιο αυστηρές οξύτερες και πιο αποτελεσματικές. Δεν κάνουν μόνο λόγο για την διατήρηση απλώς κάποιων κυρώσεων, αλλά για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους. Αν δει λοιπόν τώρα κανείς τι κάνει, τι πράττει η Ρωσία, τίποτα το καινούριο ξεχωριστό δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν καλά μαντάτα δηλαδή και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε εδώ και να το λάβουμε υπόψη. Και ας θυμόμαστε πάλι επίσης ότι η συμφωνία Μίνσκ 2 δεν αναφέρει καν την Κρυμαία, δεν αναφέρει καν το θέμα επιστροφής της. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση που συζητάμε πιστεύω είναι άριστη διότι είναι ακριβής είναι ακριβής και αυστηρή γιατί δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει η κατάσταση. Είδατε στο ντοκιματέρ ότι αναφέρθηκε ότι είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα και τώρα ε, αυτά, για την κρίση της Κρυμαίας και τώρα είπαν ε, για τη Δανία ότι μπορεί τα πλοία της να αποτελέσουν στόχους. Είναι όχι απλά δύσκολη η κατάσταση, είναι ανεύθυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας. Δεν μπορεί να καθίσει κανείς με τον κύριο Πούτιν και να συζητήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Πούτιν είναι να εφαρμόσει τη Συμφωνία Μίνσκ 2. Να κάνει δηλαδή αυτά που υποσχέθηκε και που θεσμεύτηκε να κάνει. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εχθροί της Ρωσίας ή των Ρώσων. Οπότε σε αυτή την έκθεση και θα δούμε τι μορφή θα λάβει όταν τροποποιηθεί και όταν θα την ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Ε, πρέπει να εστιαστούμε και σε αυτό στη συνεργασία με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που θέλουν να κάνουν τη Ρωσία πιο δημοκρατική, να συνεργαστούμε με τους φοιτητέ, γιατί δεν είμαστε εχθροί του ρωσικού λαού. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και δεν είναι business as usual το να απειλεί κανείς με πυρηνικά όπλα. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει κάθε λογικής. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σόλτς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την κατάθεση αυτού του σχεδίου. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει από την άλλη πλευρά με τον τρόπο που θα έπρεπε. Πιστεύω πρέπει να προβληματιστούμε σε βάθος. Γιατί το 2005 το 2015 και μάλιστα την άνοιξη 2015 όταν είχαμε και τις, ε, ε, ε τις ε, για τα 70 χρόνια από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με τη στρατηγική εταιρική σχέση που τα τελευταία χρόνια τη σχέση με την Ρωσική Ομοσπονδία οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και να δούμε και να αναλύσουμε τα πράγματα και να το πούμε εδώ ειλικρινά. Πρόκειται για καλές γειτονικές διμερείς ομαλές σχέσεις που με τη Ρωσία πρέπει να αναπτύσσονται και όχι κατά της Ρωσίας. Διότι κατά της Ρωσίας δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά λοιπόν, στρατηγικές θέσεις ε, που εισάγονται εδώ. Πρόκειται για τα θέματα οικουμενικής εμβέλειας εδώ, παγκόσμιας ε, εμβέλειας. Η κυρία Γιακονσάρη το ανέφερε. Πρόκειται για τις κοινωνικές αντιφάσεις στην ίδια τη Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ακροδεξιά κόμματα ε, και έχουμε και ε, δεξιούς που συνεργάζονται και όταν βλέπουμε αντίστοιχες τάσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και τι είναι προς το συμφέρον μας. Και το αναφέρω αυτό συνειδητά πρόεδρε. Όταν θα ήθελα να πω ότι ο Στούρμα γράφει στην εφημερίδα Βέρτ το Σαββατοκύριακο η Δύση είχε συμπεριλάβει λέει την ε, Ρωσία στο παγκόσμιο σύστημα στην Δύση πρέπει τώρα να θέσουμε το εξή ερώτημα. Τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα, πώς θα διαμορφωθεί η σχέση με τη Ρωσία για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τι θα γίνει σε σχέση με τον εξυγχρονισμό της εταιρική σχέσης. Νομίζω σωστές ερωτήσεις διαπιστώνει ο κύριος Τούρμερ στην εφημερίδα Welt. Πρέπει να καταστήσουμε σαφέστερο πώς με τις διεθνείς αυτές προκλήσεις στην εταιρική σχέση με τους Ρώσους θα προχωρήσουμε. Έχω και πολλέ άλλε παρατηρήσει. Θα θέλω να συνεργαστούμε συνεργαστώ με τον συγητή για την ολοκληρωθεί η έκθεση όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι, ξέρετε, ότι <clears throat> δεν επιβάλλουμε σε κανένα τίποτα, δεν ε, επιβάλλουμε και δεν κάνουμε καμιά εισβολή σε κανέναν εμείς. Άρα λοιπόν πρέπει το θέμα της Ρωσίας να εξεταστεί ξεχωριστά. Εσείς έχετε το λόγο για δύο λεπτά δεν θα χρειαστώ και αυτά τα δύο λεπτά ο κύριος Μέζεριτς. Θα έπρεπε να εξεταστεί και να συζητηθεί αυτή η έκθεση και θα θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Λαντσμπέργκη στον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε για αυτή την έκθεση. Είναι πραγματικά η έκθεση ε, οξία σε κάποια σημεία, σε άλλα σημεία όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για μια έκθεση αυτού του χαρακτήρα. Είναι κάποια στοιχεία όμως όπου εμείς θα θέλαμε κάπως διαφορετικές θέσεις να εκφράσουμε. Γι' αυτό προσβλέπουμε στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι ο μόνος τρόπος να επιληθούν τα προβλήματα είναι με μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινή πολιτική και πολιτικές που θα εφαρμόζονται με ένα συνεκτικό και ε, συνεπή τρόπο. Ο λόγος για τον οποίο διαφωνούμε για τα γεγονότα του 2008 είναι για το ότι δεν ήταν η Ευρώπη η οποία επέστρεψε στις κανονικές εργασίες της, αλλά τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Δεν είναι λοιπόν, ας το πω έτσι, κάποια αφηρημένη έννοια ή ένα γενικό όργανο Ευρώπη που άλλαξε πολιτική. Τα κράτη-μέλη, αν θέλουμε να αποφύγουμε να επαναληφθεί αυτό, χρειάζεται μια ισχυρότερη κοινή εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα σημείο του οποίου λοιπόν υπάρχει συμφωνία η έκθεση κάτι θα πρέπει να πει για τους μακροπρόθεσμους στόχους έναντι της Ρωσίας και είναι σημαντικό να αναφέρει τη μακροπρόθεσμη συνεργασία με τη Ρωσία και θεωρώ ότι η συνεργασία με τη Ρωσία είναι αναγκαία αλλά και εφικτή, δυνατή και μια ολόκληρη σειρά προϋποθέσεων προαπαιτουμένων που χρειάζονται είναι και η επιστροφή στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η κατάσταση ε, όσον αφορά την Ρωσία, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και αλλού, έχει ε, πάρει ε, κρίσιμες διαστάσεις, είναι κέρια σημασία όλα αυτά, αλλά πάλι δεν έχουμε ακόμα τον ψυχρό πόλεμο. Υπάρχει μια δυνατότητα να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Καστάντο, δύο λεπτά παρακαλώ. Δεν παρίσταται, πολύ καλά. Ο κύριος Κέλλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Λαντσπέργκερ, γιατί τέτοιες εκθέσεις τις χρειαζόμαστε. Και όπως πολύ σωστά μας είπε, δεν πρόκειται για το ότι θέλουμε να ακολουθούμε την επικαιρότητα και να αλλάζουμε κάθε τόσο. Η έκθεση αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει μια αξιολόγηση επί της αρχής και δεν πρόκειται μόνο για τους Ρώσους, δεν έχουμε καμία εχθρότητα απέναντι στους Ρώσους αυτούς καθ' αυτούς, είναι θέμα συμπεριφοράς της ρωσικής ηγεσία. Αυτή είναι η οποία θυμίζει συνέχεια από την εποχή τη Σοβιετική, της ΚΑΚΕΜΠΕ. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα είναι ενότητα και θάρρος απέναντι σε θετικές αντιδράσεις γιατί βλέπετε δεν αντιδράσαμε σοβαρά νωρίτερα για αντίστοιχε ε, τέτοιες παραβιάσεις ε, διεθνούς δικαίου όπως ήταν ε, η περίπτωση της εισβολής στη Γεωργία. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτά που κάνει στην Ουκρανία. Αλλιώς η επίθεση αυτή θα ξαπλωθεί και θα μας υπεράσει όλους. Ο Υπουργός της Εστονίας που ήταν εδώ τις προάλλες είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο Β της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Αναφέρθηκε στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία αναφέρθηκε επίσης στην, στις προμήθειες όπλων. Πάντως, ό,τι δισταγμούς έχουμε σήμερα, εφόσον δεν υπάρχουν θετικά μηνύματα από τη Ρωσία, θα σήμαινε ότι όσα γίνονται, γίνονται σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Θέλω να αναφερθώ όλους ιδιαίτερως στην παράγραφο 10, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική σήμερα που μιλάει για έναν θετικό μηχανισμό αντιμετώπισης της ρωσικής προπαγάνδας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, επί της αρχής πάντα υπάρχει ένα σχέδιο Β, δηλαδή δηλώνουμε ότι νικήσαμε και επιστρέφουμε στη χώρα μας. Ο κύριος Μαμικίνης τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Ο κύριος Λαντσβέργης ετοιμάζει μια έκθεση που όλοι περιμένουμε. Βέβαια είναι πολύ ατυχές το πλαίσιο μέσα στο οποίο ετοιμάζεται η έκθεση αυτή. Χτες εγκρίναμε ένα ψήφισμα και είχαμε έναν εκπρόσωπο. Τώρα έχουμε την έκθεση αυτή, εγώ διαβάζω την έκθεση και βλέπω ότι τελικά πρόκειται για το ίδιο κείμενο, η ίδια διατύπωση, ξανά και ξανά τα ίδια. Τίποτα καινούριο. Οπότε εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται αυτή η έκθεση. Για να επηρεάσει τη Ρωσία. Οι Ρώσοι έχουν ε, αναπτύξει ανοσία σε τέτοιου είδους εκθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούνε σαν σημάδια δυναμίας από τη δικιά μας την πλευρά. Δεν πρόκειται εξάλλου να πείσουμε όλους τους ευρωβουλευτές ή την Επιτροπή να κάνει κάτι παραπάνω. Φοβάμαι δηλαδή ότι κάθε έκθεση που ετοιμάζουμε έχει τέτοια ισχύ ώστε τελικά μας αποδυναμώνει όσο περνάει ο χρόνος. Και εδώ κινδυνεύουμε να πέσουμε σε λόγια και όχι πράξεις πάλι θα είναι κάτι σαν σπαμ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι οι επαφές μεταξύ ατόμων, διπλωματία μεταξύ ανθρώπων. Ακούσαμε και πριν μια πρόταση. Υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τη Ρωσία. Για παράδειγμα, Ιράκ. Το συζητήσαμε πριν από λίγο. Συνεπώς, κάποια βήματα μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, αλλά αν οι Ρώσοι δεν θέλουν να ακούσουν ότι σφάλουν, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να τους το λέμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να το λέμε. Ο κύριος Τάνοκ τώρα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λαντσπέργκης αλλά και να ζητήσω συγγνώμη στον παππού σα ο πριν από 10 χρόνια όταν τον πρώτο συνάντησα μα προειδοποιούσε διαρκώ για του κινδύνου ε, που θα παρουσίασε στο μέλλον η Ρωσία και εγώ ήμουν ε, ε, αναπληρωτή συντονιστή σε εκείνη την ομάδα τότε και τον αγνόησα. Αλλά είχε δίκιο και εγώ είχα άδικο και το παραδέχομαι. Και αν παρακαλώ δείτε τον παππού σας που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μεταφέρετε του τη συγγνώμη μου. Ε, τα όσα ισχυριζόταν τότε βρίσκονται εδώ σε αυτή την έκθεση και την υποστηρίζουμε όπως είπαμε και ε, αυτή την εποχή στις χώρες σας ε, θα πρέπει να φροντίσετε, να μεριμνήσετε ώστε οι στρατοί σας να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τυχόν επίθεση της Ρωσίας. Ε, επίσης αυτή την εβδομάδα η άκρα δεξιά, τα άκρα δεξιά κόμματα και το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας αρνείται να συμμετάσχει στις συναντήσεις αυτές ε, ε, ε, και συμμετείχε συναντήσει στο Πίτερσμπουργκ, στην Μετρούπολη, όπου εκφράζεται η υποστήριξη προς τη Ρωσία. Είπε κάποιος ότι ο καθένας φαίνεται από τους φίλους του, φαίνεται ότι είναι από τους φίλους του. Είναι ένα φασιστικό ε, κόμμα σήμερα, μια ε, φασιστική κυβέρνηση που βρίσκει στήριξη αυτή τη στιγμή στο ε, Πετρούπολη και και τα δικά μας ακροδεξιά κόμματα προσπαθούν να γίνουν φίλοι με τους Ρώσους Έχω μια ερώτηση για την παράγραφο 2. Έχω πει επανειλημμένω ε, προσωπικά ότι μια στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, δεδομένη των επιθέσεων και των παραβιάσεών τη, ε, ε, πρέπει να σταματήσει. Ποια διαδικασία υπάρχει για να σταματήσουμε τη στρατηγική συνεργασία. Χρειάζεται ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο. Μπορεί Μπορούν τα κράτη-μέλη να πούν δεν θέλουμε πια αυτή τη στρατηγική σχέση. Πώ τη τερματίζουμε, δεν το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζω, και τέλο θα ήθελα να θυμίσω τα εξωφρενικά σχόλια του Ρώσου πρέσβη στη Δανία που απειλεί με το ναυτικό τους ε, ως στόχος πυρηνικών όπλων. Είναι κάτι εντελώς ανεύθυνο. Ε, είναι χειρότερο από ό,τι είχαμε ακούσει και για τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για να σου πω την αλήθεια. Ε, ευχαριστώ, κύριε Ραστριβίτσιος, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον Καμπριέλη για τις ε, προσπάθειες του για αυτή την έκθεση για τη Ρωσία και πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να ακούσουμε. Τι κείμενο θέλουμε να έχουμε. Η κατάσταση στη Ρωσία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ακούσαμε απαράδεκτα σχόλια από Ρώσους εξωματούχους πρόσφατα και να μην ξεχνάμε την πρόσφατη συνθήκη μεταξύ Ρωσίας ε, ε, που σημαίνει προσάρτηση και κατάληψη την ε, συνάντηση νεοναζί και φασιστών πρόσφατα στο Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη είχε υποφέρει για 900 μέρες ε, από τους Ναζί η Αγία και τώρα έχουν ξαναεπιστρέψει. Το μόνο μέλος της Ντούμα που καταψήφισε την προσάρτηση της Κρεμαίας ε, δεν επιτρέπεται τώρα να επιστρέψει στη Ρωσία και είναι πρόσφυγα στις ΗΠΑ. Συνάδελφοι, ας μην φοβόμαστε τις κόκκινες γραμμές. Δεν αναμένω κάποιο δικό χάρτη για το πώς πρέπει να εξελίξουμε τώρα τη σχέση μας με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει τέτοια διάνοια στον κόσμο για να το λύσει αυτό. Η απάντηση βρίσκεται στο Κρεμλίνο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ ε, και τι θα επιβάλλουμε ω κύριο στη Ρωσία. Θα ήθελα μάλιστα να τονίζουμε περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου η κατάσταση είναι φρικτή και επιδεινώνεται διαρκώ. Όπω και η κατάσταση των γειτονικών χωρών που ε, δεν, που τους, δεν, δεν επιτρέπεται η ελεύθερη επιλογή για ένα ευρωπαϊκό μέλλον από το Κρεμλίνο. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και εύχομαι να συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία μέχρι το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καστάλντο επέστρεψε, μπορεί να έχει το λόγο για δύο λεπτά και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον εισηγητή είναι σημαντικό να κάνουμε και κάποια αυτοκριτική σε αυτή την έκθεση. Παρότι φυσικά έχει τεράστιες ευθύνε ε, η Ρωσία για αυτή την κρίση, αναρωτιέμαι το εξή. Κάναμε εμείς ό,τι μπορούσαμε πριν από ένα χρόνο και σήμερα για να αποτρέψουμε ε, περαιτέρω επιδείνωση. Προηγουμένως μιλήσατε για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη που θα βγει από αυτή την κρίση επικεντρωνόμενος ε, στην προπαγάνδα και στον ενεργειακό πόλεμο και θέλω να σας ρωτήσω είστε σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει πιο ε, ισχυρή από ένα τέτοιο ενεργειακό πόλεμο. Αν υπήρχε τέτοιο πόλεμο, ε, θα είχαμε χάσει, πιστεύω, πριν καν ξεκινήσει. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Να επενδύσουμε δηλαδή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση, στη μείωση τη κατανάλωση ώστε να έχουμε μεγαλύτερη όντως αντοχή σε σχέση με την εισαγωγή δρομοναθράκων από την οποία εξαρτώμαστε ε, δεδομένης και της ε, ταυτόχρονης κρίσης με τη Λιβύη. Ε, και ειλικρινά τώρα όσον αφορά το άνοιγμα προς το διάλογο, ναι σύμφωνο, η διπλωματική οδός είναι κατά την άποψή μου είναι ίσως όχι η καλύτερη αλλά είμαι πεπισμένο ότι είναι η μόνη δυνατή λύση και η μόνη εφικτή. Προσωπικά θα ήθελα να αποφύγουμε ε, πράγματα όπως αυτά που αναφέρατε. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε μια διπλωματική διαπραγμάτευση ε, με το σκεπτικό ότι πρέπει να τους διδάξουμε ε, κάποιο μάθημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να κρίνουμε και τους εαυτούς μας και αυτούς, αλλά να έχουμε έναν ε, ε, ανοιχτό διάλογο και όχι σύγκρουση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Κύριε Πλένκοβιτς, έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πάσκο. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον φίλο μας ε, Γκαμπριέλος Λαντσπέργκης. Είναι εξαιρετική, πιστεύω, η έκθεσή του. Θα τη συζητήσουμε μέσα στι επόμενες εβδομάδες. Η μόνη πτυχή που μάλλον λείπει είναι κάποια εμβάθυνση, επειδή αναφέρεται στον τίτλο «Κατάσταση των σχέσεων» μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Αλλά από όσο κατάλαβα, αυτό ε, μπει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής τα περισσότερα. Συμφωνώ με τους περισσότερους συναδέλφους, υπάρχει κάτι που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που θέλει να δώσει ο εισηγητής, είναι η αλληλεγγύη και η ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Αυτή πιστεύω είναι η σημαντικότερη γραμμή αυτού του εγγράφου που το καθιστά εντελώ διαφορετικό από τις προηγούμενες παλιότερες εκθέσεις για τη Ρωσία και είδαμε τώρα ε, και στο παράδειγμα στην περίπτωση της Ουκρανίας ε, και στο, ε, στην περίπτωση άλλων ε, γειτονικών χωρών όπου ενορχιστρώνονται διενέξεις από τη Μόσχα ε, και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε σε μια τέτοια πολιτική. Πιστεύω επίσης και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκινήσουμε άμεσο, έμεσο ε, διάλογο, να υποκινήσουμε κάποιες άμεσες, έμεσες ε, αλλαγές στη ρωσική κοινωνία και να υποστηρίξουμε τις αλλαγές που θα οδηγήσουν τη Ρωσία σε μια πιο πλουραλιστική και δημοκρατική οδό, θα αποδεχθεί τις αξίες που διακατέχουν ε, την πολιτική συνεργασία στους διάφορου τομεί. Ε, Καλώς ορίζω λοιπόν τι τροπολογίε και περαιτέρω συζητήσεις επί τη εκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιουρέκ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ κι εγώ τον εισηγητή. Είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για μελλοντικές συζητήσεις. Η έκθεση αυτή μάλιστα αξίζει ακόμα περισσότερο επειδή την ε, εκπονεί κάποιος που προέρχεται από μια χώρα που συνορεύει με την ε, Ρωσία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί ως κάτι επιπλέον σημαντικό. Κάτι όμως λείπει εδώ. Ξέρουμε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν πολύ προπαγάνδα απέναντι της Ευρώπης. Λένε ότι μας ε, επιτίθενται ναζιστές, φασιστές. Η Ρωσία έφτασε να προτείνει στα Ηνωμένα Έθνη ψήφισμα κατά της προσπάθειας που γίνεται κάποιοι να μιλήσουν κατά του κομμουνιστικού παρελθόντος της. Υπάρχουν όμως και Ρώσοι που θέλουν να γνωρίζουν την αλήθεια για τα θύματα του σταλινισμού, του κομμουνισμού, του κομμουνιστικού καθεστώτος δηλαδή της εποχής εκείνης. Ας θυμόμαστε το εξή. Όταν ο Πούτιν λέει ότι κάποιος προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αυτό που εννοεί είναι ότι εκείνος θα ήθελε να μιλάμε υπέρ του Στάλιν, να γράψουμε θετικά πράγματα για την κομμουνιστική περίοδο. Ο κομμουνισμός δεν έχει να κάνει μόνο με επιθέσεις στη δεκαετία του 30 του 40 ή όταν ε, έγιναν επιθέσεις στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, πρόκειται και για τη δεκαετία του 70 και για τις προσπάθειες που έκανε η Σοβιετική Ένωση τότε. Εμείς καταδικάζουμε το κομμουνισμό διεθνώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ηθική τάξη. Εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια όσον αφορά τη Ρωσία. Βλέπουμε τι σύστημα θέλουν να επαναφέρουν στη Ρωσία. Πρόεδρος, λέτε ότι κάποιοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία, <laughs> κάποιοι θέλουν να την ξαναφτιάξουν όμως. Ο κύριος Μπουτικόφ τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ έχει πει ότι μπορείτε στα λόγια να είσαστε ήπιοι, αλλά σκατάτε και ένα ραβδί καλού κακού. Εγώ νομίζω ότι το σχέδιο αυτό έκθεσης είναι θύμα της υπόθεση ότι και το αντίθετο είναι αλήθεια. Ότι δηλαδή αν δεν τα καταφέρνεις με το ραβδί, ας έχεις σκληρό λόγο. Εγώ είμαι κατά μια τέτοια τάση, ιδιαίτερα όσον αφορά την προτινόμενη παράγραφο 4 της έκθεσης αυτής. Η παράγραφος αυτή μιλάει για διάλογο, ότι ως προϋπόθεση πρέπει να έρθει ο διάλογος. Μα ο διάλογος δεν είναι το εναλλακτικό. Δεν είναι εναλλακτική λύση αντί να έχουμε κυρώσεις να έχουμε διάλογο. Όχι. Αν όμως πιστεύουμε ότι ο διάλογος είναι αναγκαίος, το να βάζουμε προϋποθέσεις για διάλογο, αυτό είναι κάτι που θα δυσκολεύσει το διάλογο. Θέλουμε διάλογο ειρήνης με τους Παλαιστίνιους, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να το κάνουμε σαν να μην υπάρχει τρομοκρατία και μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη τρομοκρατία χωρίς να υπάρχει ειρηνικός διάλογος. Δεν είναι σωστή προσέγγιση εδώ για προϋποθέσεις στο διάλογο. Και στις επόμενες προτάσεις τι λέει, λέει ότι ο διάλογος πρέπει να αρχίσει και πάλι μόνο εφόσον προηγουμένως έχουμε πετύχει να επιστραφεί η Κρυμαία στην Ουκρανία. Αυτή είναι η προϋπόθεση για το διάλογο δηλαδή. Δηλαδή αναβάλουμε το διάλογο για και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα. Σωστό είναι αυτό πολιτικό. Θα ήταν σωστό να λέγαμε, επειδή δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξει επανένωση της Γερμανίας, γι' αυτό δεν μιλάμε με την άλλη πλευρά, θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο. Με αυτό μας φέρνει σε αδιέξοδο μια τέτοια προσέγγιση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Βάτρανς τώρα. Και έπρεπε να είχε πάρει το λόγο πριν από τον κύριο Πατικόφερ, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δύο λεπτά. Κανένα πρόβλημα, Πρόεδρε λέει η κυρία Βάτμενς, θα μιλήσω φλαμανδικά, γιατί είναι πιο εύκολο για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, εισηγητή για τα σχόλιά του. Τελικά είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να μιλήσουμε. Είπαν και οι συνάδελφοι ότι κάθε μέρα περνάει ανταλλάσσουμε απόψεις. Η έκθεση αυτή, τη διάβασα εγώ τουλάχιστον στα Ολλανδικά και κάπου υπάρχει σκληρή γλώσσα. Υπάρχουν δύο σημεία όμως που πιστεύω εγώ ότι δεν έχουμε και θα ήθελα να προσθεθούν. Το θέμα της προϋπόθεσης για το διάλογο και το θέμα της επικοινωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι στα σύνορα της Ευρώπης και ότι ένας γείτονας παραμένει πάντα γείτονας. Γι' αυτό καλό θα ήταν να μπορούμε να προσθέσουμε κάτι όσον αφορά για το πώς βλέπουμε το μέλλον. Είδαμε η Μογκερίνη στο Στρασβούργο τι μας είπε πρέπει να το σκεφτούμε αυτό ξανά και ξανά είπα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφοροι νέοι Ρώσοι οι οποίοι έχουν πολύ αρνητική εικόνα για την Ευρώπη. Αυτή η γενιά θα είναι η επόμενη ηγεσία της Ρωσίας. Ε, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος μας στην Ρωσία. Το δεύτερο που θα ήθελα να προσθέσουμε είναι κάτι για τις οικονομικές συνομιλίες και πόσο κοστίζει στην Ευρώπη το μποϊκότ που κάνει η Ρωσία στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Γνωρίζετε βέβαια ότι κάποιοι από εμά είμαστε πιο γείτονε με τη Ρωσία από ότι κάποιοι άλλοι. Και να ξέρετε ότι εμείς δεν ε, κάνουμε προπαγάνδα στους νέους εναντίον της Ευρώπης. Εκείνοι το κάνουν, ό,τι και να κάνουμε εμείς. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κύριος Κάρλουρ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Για την αναγνώριση των προβλημάτων σε σχέση με τα κράτη υπό ένταξη, όταν υπάρχουν έντονα τέτοια αισθήματα για το ότι ο κύριος Πούτιν δεν είναι ίσως ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άτομο. Αλλά να δούμε επίσης τι γίνεται ότι βρίσκεται ο Πούτιν σε μια θέση που θέλει να δείξει ότι έχει μια στεναρή θέση να αποδείξει στους Ρώσους ότι είναι ο ισχυρός ανήρ και αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία και σε σχέση με την, ε, ε, το εβραϊκό, ας το πω έτσι, τις εβραϊκές ε, προεκτάσεις. Αυτό που είδαμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί μια πιο φεντεραλιστική τάση. Και θα δούμε ότι εδώ τονίζεται σωστά ότι Υπάρχει η τοποθέτηση από διάφορους ε, πολιτικούς ε, στο εύρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι εδώ αφήνουμε, επιτρέπουμε να υπάρχει περισσότερη ομοσπονδιακή τάση και κίνηση και αυτό σε σχέση με την, τις δαπάνες για την άμυνα δημιουργεί μείζον πρόβλημα σε σχέση με τα περισσότερα κράτη-μέλη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ευκαιρία όπως τονίστηκε και από τον κύριο Γιούγκερ πρόσφατα, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπομειστεί τις ευθύνες της. Μια διπλωματική πρωτοβουλία είναι η μόνη όμως εναλλακτική λύση παρότι θα ήθελαν κάποιοι να δείξουν μια στεναρή στάση. Πρέπει όμως να υπάρξει η δυνατότητα να έχουμε επαφές για να επιληθούν τα προβλήματα. Εξίσου πρέπει, έπρεπε δυστυχώς το 1940 να έχουμε σχέσεις και επαφές με τον ε, Στάλιν για να ε, καταπολεμηθεί η ε, ναζιστική απειλή. Το ίδιο λοιπόν εδώ πρέπει να ισχύει σε σχέση με το σημερινό σκηνικό. Θα πρέπει να δούμε σε σχέση με την τάση αυτή που ακολουθήθηκε τότε το 1930 και σήμερα και σε σχέση με την απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε μεγαλύτερη τέτοια βούληση. Ο κύριος Μποργέτσιο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλες τις ιστορικές αναφορές που θεωρούν απαραίτητο να αναφέρουν πολλοί συναδελφοί. Ως ε, ιδεολογία που πρέπει να ακολουθούμε. Εγώ ανήκω στη γενιά που έζησε και συμμετείχε όσο ήταν δυνατόν ε, στον αγώνα απελευθέρωσης ε, της ε, Ανατολής της Ευρώπης από τον κομμουνιστικό πολιταρχισμό. Θυμάμαι εκείνη την εποχή ελάχιστοι ήμασταν που σηκώσαμε τη σημαία της ελευθερίας. Ήμασταν οι ελάχιστοι νέοι που πηγαίναμε να ε, μοιράσουμε προκηρύξει στην κόκκινη πλατεία. Όλοι οι υπόλοιποι κάθονταν σπίτι τους ήσυχα και έκαναν εμπόριο με τη Σοβιετική Ένωση. Και τώρα βλέπω ότι όλοι έχουν συνταχθεί κατά αυτού του θανάσιμου εχθρού της ελευθερίας και της ε, Ευρώπης που είναι ο Πούτιν στη Ρωσία. Και βλέπω ένα έγγραφο σαν αυτό που μου φαίνεται περισσότερο ως ανάκριση παρά ως ε, πολιτική πράξη που εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας Ευρώπης που θέλει την ειρήνη. Ξέρετε, οι λαοί μας θέλουν ειρήνη. Το ξεχνάμε αυτό το επιχείρημα. Θέλουν να δουν πώς ε, μέσω κάποιου διαλόγου, χωρίς παραχωρήσεις, διαλόγου από θέση ισχύω, χωρί όμω ε, ιδεολογικέ προκαταλήψει. Το έγγραφο αυτό πρέπει να το πετάξουμε στα σκουπίδια, διότι έχει μια λάθο προσέγγιση πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών μας και όχι ξένα συμφέροντα. Όταν η Ευρώπη βρισκόταν υπό τον ζυγό ε, μιας απολυταρχίας η Σοβιετική, όπως η Σοβιετική Ένωση ξεχάσαμε να σηκώσουμε τη σημαία της ελευθερίας γιατί τότε κάναμε εμπόριο μαζί τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι, εκείνη την εποχή ήταν αγώνας για την ειρήνα, ε, από όσο λέγαμε. Ε, λοιπόν, κύριε Λαντσμπέργκης, ε, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συναδέλφοι για όλα τα σχόλια. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε φυσικά τη συζήτηση και στο μέλλον και πολλά από αυτά που θα πούμε και που είπαμε εδώ πέρα θα ε, συμπεριληφθούν στη τελική μορφή της έκθεσης. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω, όπως αναφέρονται πολλοί, υπάρχει μια βάση συνεργασίες ε, και μια βάση για μη συνεργασία. Κάποιοι από σας είπατε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε ή να ξεκινήσουμε να συζητάμε και γενικώ να συζητάμε. Ξέρετε, το έχουμε ήδη κάνει αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο να συζητήσουμε. Εμείς ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Όλοι μας. Το πρόβλημα είναι από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, δεν συζητάμε γιατί εμείς κάνουμε κάτι λάθος και μετά παραμένουμε σιωπηλοί και αρνούμαστε να μιλήσουμε. Πώς να μιλήσουμε μετά από τη θαλατηφόρο, από τη, από τη μοιραία πτήση ε, της Malaysian Airlines, την πτήση 17. Τι να συζητούσαμε τότε. Τι έπρεπε να συζητήσουμε αν καταλάβουν τη Μαριούπολη. Εντάξει, δεν μας συμφέρει να παραμένουμε σούπηροι. Πρέπει να μιλάμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν με διασκεδάζει λοιπόν καθόλου το να μου λέτε ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διάλογο υπό προποθέσει. Πρέπει να είναι υπό προποθέσει. Όταν σκοτώνουν ανθρώπου στον δρόμο με εντολέ από το Κρεμλίνο, δεν μπορούμε εύλογα να λέμε ότι θα συζητάμε χωρί προποθέσει. Και μια σύντομη δήλωση για να ολοκλώσω. Εάν ο κύριο Πούτιν σταματήσει το σοβαρό πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώ κάτι θα του προσφέρει η Ευρώπη. Ε, κάτι για τα γαλακτοκομικά ή κάποια ευκολία κάτι τέτοιο. Εάν ο κύριος Πούτιν συνεχίσει και καταλάβει τη Μαριούπολη, τότε θα υιοθετήσουμε σκληρή θέση, θα ακολουθήσουν χειρότερες κυρώσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια κοινή λύση τώρα, η οποία θα χαρακτηρίσει την ε, στρατηγική στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο η πρώτη μου πρόταση είναι να σκεφτούμε τα όσα συνέβησαν, στα 19 χρόνια των σχέσεων μεταξύ μας και να αναγνωρίσουμε ότι οι κόκκινες γραμμές του διεθνούς δικαίου υπάρχουν και ότι έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη και θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για να ξανακολλήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να επενθυμίσω ότι Δευτέρα 30 Μαρτίου στι 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για τι τροπολογίε. Πρέπει να σα ανακοινώσω ότι το Κοινοβούλιο θα κλείσει τι πόρτε του Αμέσω μετά Οπότε αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία, δεν υπάρχει δυνατότητα παράταση. Και τώρα να σα ευχαριστήσω και να καλέσω τον συνάδελφο τον κύριο Πλένκοβιτς να έρθει να προεδρεύσει. Ευχαριστώ πολύ Αντιπρόεδρε Πάσκο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με το σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Πρώτα θα δούμε τα σκεπτικά και μετά τον ρόλο της ε, Επιτροπής Εξωτερικών σε σχέση με την ανακοίνωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια και η Επιτροπή Ήτρε θα ψηφίσει τον Απρίλιο από αυτού του εγγράφου. 52 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν και κατέθεσαν προτάσεις και τους κοιόδης εισηγητές και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς άρρηκτα αποτελεί τμήμα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι οι ενεργειακοί πόροι χρησιμοποιούνται περισσότερο κάθε φορά ως μέσο και εργαλείο για την εξωτερική πολιτική και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλήγματα εξωτερικής προέλευσης όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Και αυτά έχουν άμεση επίπτωση και επενέργειες στην καθημερινή μας ζωή. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή συνάδελφο Άρνε Λίτσε που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ θερμά Πρόεδρε. Την κατάσταση την περιγράψατε ότι σε σχέση με την Επιτροπή Πολιτισμού που θα έχουμε κοινή συνεδρίαση πιέζει ο χρόνος και θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να προσθέσω τη φωνή μου και να εκφράσω ευχαριστίες προς όλους που συμμετείχαν για την συνεργασία τους. Να ευχαριστήσω λοιπόν οι σκιώδεις εισηγητές πολύ καλά συμμετείχαν χρονικά σε αυτή την αλληλουχία και με τις τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες ώστε οι περισσότερες τροπολογίες να μπορέσουν να συγχωνευτούν σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Το σημαντικότερο έργο για μας για την εξωτερική πολιτική είναι να δούμε τις διεθνείς επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε συζήτηση με τη Ρωσία καταδεικνύεται πόσο είναι σημαντική μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και αυτό το έγγραφο αφορά την τοποθέτηση, τοποθέτηση ρητά το αναφέρω, της δικής μας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδότηση σε σχέση με ενεργειακά προϊόντα. Μια και πιέζει ο χρόνος δεν θα υπησέθω σε θέματα ε, ουσίας αν έχουν κάποιοι παρατηρήσεις ε, θα μπορούσα να το έκανα. Θέλω να αφήσω το χρόνο για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιοι από τους σκιώδεις εισηγητές θα ήθελαν ίσως να παρέμβουν, να παρουσιάσουν κάποιες δικές τους σκέψεις, να ληφθούν υπόψη. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λοιπόν προτείνω να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε. Λοιπόν, πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν και αρχίζουμε την ψηφο, τις με τις ψηφοφορίες. Έχουμε τον πρώτο συμβιβασμό, συμβιβασμό 1. Ποιοι είναι υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6, επειδή άλλες έχουν καταπέσει. Ποιοι είναι υπέρ της 6. Κατά. Άποχες. Απορρίφθηκε η τροπολογία 6. Συμβασμός 2 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 22, υπέρ της 22, κατά, άποχες, απορρίφθηκε. Τροπολογία 23, υπέρ, κατά, άποχες, Απορρίφθηκε. Τοπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ήθελα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 35, άρχεται η ψηφοφορία. Μια στιγμή. Εντάξει λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 28 εναντίον, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 4 τώρα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 5 υπέρ αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε στις ε, ατομικές επιμέρους τροπολογίες. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Τροπολογία 51 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. 52 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία εν τέλει 6 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και τελική τώρα ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά όμως, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 39 υπέρ 9 εναντίον 3 αποχης αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον συνάδελφο κύριο Λίτς. Εγκρίθηκε η γνωμοδόση, υιοθετήθηκε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 5.30 όπου θα ξεκινήσει η κοινή συνεδρίασή μας με την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ.